Πιστεύουμε, τρίτο, ότι μια περαιτέρω εξέλιξη της ρύθμισης για το κόστος και τους κινδύνους είναι δυνατόν αυτά να μειωθούν. Πρόκειται για 200 δισεκατομμύρια για τα επόμενα 10 χρόνια. Εγώ ανισχόλου και περισσότερο για το γεγονός ότι στον τομέα της ενέργειας από την έρευνα μέχρι την παραγωγή, μέχρι την υποδομή, μέχρι την αποθήκευση, μέχρι την εξοικονόμηση ενέργειας Εκεί λοιπόν σε όλους αυτούς τους τομείς δαπανώνται υπερβολικά λίγα χρήματα. Και τα κίνητρα, αλλά και η ασφάλεια σχεδιασμού, η διαφάνεια. Από πλευράς ενεργειακής πολιτικής που απευθύνεται στους επενδυτές δεν είναι αρκετά ελκυστική. Γι' αυτό λοιπόν η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου μέσω της ΕΙΣΑ μέσω των εθνικών ρυθμιστών με αναλύσεις κόστους-οφέλους με έντιμες αποζημιώσεις για μένα μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Και τέταρτο, η ενδεχόμενη κατά περίπτωση συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 50-60% όλων των έργων δεν θα χρειαστούν καν συγχρηματοδότηση πολλά έργα θα χρειαστούν μια μικρή συγχρηματοδότηση. 10, ίσως λίγο παραπάνω της 100. Αλλά από την εμπειρία των έργων που έχουμε κάνει με το EAPR, ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ένα μέρος των μέτρων που είναι απαραίτητα για την ενεργειακή μας πολιτική και που έχουν κοινό και είναι κοινού ενδιαφέροντος δεν θα χρηματοδοτηθούν από τις αγορές. Για παράδειγμα, η ένταξη των βαλτικών χωρών για υποθαλάσσια καλώδια από τη Μάλτα στη Σικελία. για την ένταξη της Μαγιόρκα στο ισπανικό και επομένως στο ενεργειακό ευρωπαϊκό δίκτυο και μεγαλύτερη πρόκληση βέβαια θα είναι η Κύπρος διότι η Κύπρος είναι η πιο απομακρυσμένη νήσος στην περιφέρεια από το Ευρωπαϊκό Κέντρο της Αγοράς Ενέργειας. Υπάρχουν φιλόδοξα προγράμματα, τα οποία τοπογραφικά είναι φιλόδοξα και επομένως έχουν μεγάλο κόστος και εκεί η συγχρηματοδότηση έχει, παίζει και ένα κατευθυντικό ρόλο για περιφέρειες της Ευρώπης όπου κάθε χώρα μέλος θέλει ε, τερματικούς σταθμούς LNC. Εκεί μια έντιμη συγχρηματοδότηση της τάξης του 10-20% μπορεί να παίξει ένα κατευθυντικό ρόλο που να είναι σημαντικός και για μια αποτελεσματικότητα κόστους ωφέλους. Αποδοτικότητα μάλλον κόστους ωφέλους. Παρουσιάστηκε χθε λοιπόν το εργαλείο μας αυτό, Connecting Europe, και έχουμε εκείνα τα 9,2 δις που σας προτείνουμε και προσπαθούμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα της ενέργειας και στον τομέα LCT με τη συνεργασία των ε, χωρών μελών με ε, δάνεια δεσμευμένα για τα έργα αυτά με χορήγηση συγχρηματοδότησης που θα συμπληρωθούν και με άλλα οικονομικοτεχνικά μέσα. Αυτά για την ώρα. Θα ξανασυναντηθούμε τον Νοέμβριο όταν θα υπάρχει το πρόγραμμα εργασιών θα το συζητήσουμε ξανά και θα συζητήσουμε τα κέντρα βάρους του ε, μαζί σας το 2012 πλέον αλλά πολύ σύντομα θα σας υποβάλουμε ολόκληρη την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής. Σα ευχαριστούμε θερμά, Επίτροπε Τινγκέρ. Περνάμε σε ερωτήσει Και πάλι, μέχρι τι και μισή έχουμε χρόνο. Πρόκειται για τι ενεργειακέ υποδομέ. Μόνο για τι πληροφορίες για αυτό το θέμα. Θα ήμουν ευγνώμων αν τώρα επικεντρωνόμασταν σε ερωτήσει επί τη ουσία. Δώδεκα έχουν ζητήσει τον λόγο. Παράκλησή μου. Ένα λεπτό καθένα ίσω. Πρέπει να το προσπαθήσουμε, παρακαλώ. Η κυρία Ντεκαστήγιο, η πρώτη, παρακαλώ. Ακολουθώντα τι συστάσεις σα Πρόεδρε. Ακολουθώντα τι συστάσει σα, Πρόεδρε. Πρώτον, Επίτροπε, συγχαρητήρια. Δεύτερον, θίξατε κέρια σημεία. Όμω το πρώτο, αυτό είναι ακόμα και πιο σημαντικό. Ο κίνδυνο, η βραδύτητα στι διοικητικέ διαδικασίε, οποιασδήποτε μορφή βραδύτητα, να αναβάλει σημαντικά και να καταστήσει πολύ λιγότερο κερδοφόρα την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών είναι πολύ υψηλός κίνδυνος παρότι έχουμε το ανώτατο των τριών ετών και την δημιουργία ενός εθνικού γραφείου που θα ελέγχει όλες τις διαργασίες. Το ξέρουμε, επειδή πολλές φορές, πολλές φορές λέω, αντιμετωπίσαμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν υπερβολικά γραφειοκρατικά βάρη και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει μια επιτήρηση, εποπτεία και μια παρακολούθηση σε σχέση με τις προθεσμίες και τα μέσα που έχουν τεθεί σχεδόν, σχεδόν καθημερινή θα έλεγα εποπτεία και φυσικά αυτονόητο είναι μόνιμη, διαρκή εποπτεία διότι σε κάποιες χώρες σίγουρα θα μπορούσαμε να δούμε προβλήματα και επιμένω σε αυτό το σημείο ιδιαίτερα διότι οπωσδήποτε θεωρώ ότι είναι κέριο μεγάλη σημασία. γι' αυτό αυτό πρέπει πρώτα να εξεταστεί ευχαριστώ Πρόεδρος ευχαριστώ Νόμπερτ Γκλάντε παρακαλώ εσείς Συγγνώμη, εσείς κυρία έχετε τον λόγο. Ευχαριστήρια, uh, Επίτροπε, και πάλι. Πραγματικά το αξιολόγησα και το εκτίμησα το ότι δόθηκαν αυτές οι επισήμασεις, Είναι πραγματιστική προσέγγιση και ευθεία. Κάνουμε λόγο για μια κρίση και πώς η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τον, το ενδεχόμενο του να κατακαιρματιστεί και πώς μπορούμε να ολοκληρώσουμε περισσότερο και να ενταχθούμε σε ένα νέο πλαίσιο περισσότερο. Δύο σημεία, δύο θέματα, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πώς στοχεύεται ή τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει για την ανάπτυξη των εθνικών ενεργειακών υποδομών, διότι αυτό είναι κάτι που χρειάζεται και δεν είναι σαφές αν τα κράτη-μέλη έχουν την πρόθεση ή τα χρήματα να αναπτύξουν τις ε, δικές τους εθνικές ενεργειακές υποδομές. Δεύτερη ερώτηση για την γενική όπως έχει η ευρωπαϊκή αγορά. Πώς αυτές οι ενεργειακές υποδομές θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος παρακαλώ. E, ευχαριστώ πολύ αξιότιμε επίτροπε. Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, θέλω και να σας ευχαριστήσω πάλι για την παρέμβασή σας και την συνεισφορά σας τα τελευταία δύο χρόνια. Εμείς κατανοούμε και αξιολογούμε το ότι τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συστήματα σαφώς με αυτή την προσέγγιση πρέπει να προσεγγιστούν και είναι σαφής η στόχη και η προσέγγιση. Και κάνω λόγο επίσης για τρίτες χώρες όλα εκείνα τα δισεκατομμύρια για τα οποία κάνατε λόγο δεν θα υπαρχέσουν με κανέναν τρόπο αυτά τα σχέδια και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είπατε οι διεργασίες, οι διαδικασίες πρέπει να επιταχυνθούν. Όμως πιστεύω ότι το θέμα θα έπρεπε, η ερώτηση θα έπρεπε να διατυπωθεί σε σχέση με την κεντρική διαμόρφωση και διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και κρατικών προμηθειών. Και σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να δούμε την κεντρική διαμόρφωση και την περισσότερο αποτελεσματική διαμόρφωση των πραγμάτων στον ενεργητικό τομέα. Ο κύριος Τούρμες. Ε, Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Τούρμες. Κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια για το ότι τις, τις υποδομές τις εγγράψατε στην ημερήσια διάταξη. Το ότι θέλετε το σχεδιασμό να τον επι, επιταχύνετε. Είναι σημαντικό να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός χωρίς η υφιστάμενη νομοθεσία για το περιβάλλον να παρακαμφθεί ή να παραβιαστεί και να μπορούν να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις νωρίτερα και να προχωρήσουν γοργότερα. Σημερίζομαι την ανάλυση σας ότι σε αυτή την χρηματοοικονομική κρίση έχουμε πρόβλημα κεφαλαίων για να βρούμε επενδύσεις και να διασφαλιστούν οι επενδύσεις όπως απαιτείται. Τρεις ερωτήσεις. Αν εμείς αυτά τα εννέα δισεκατομμύρια θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό, δεν κατανοώ γιατί θα πάρουμε μόνο ένα δισεκατομμύριο ώστε το κεφαλαιακό κόστος ε, να μπορέσει να διευκολυνθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα 8 δισεκατομμύρια τι θα τα κάνουμε. Η μόχλευση, η μοχλική επίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερη αντί ένα δισεκατομμύριο αν παίρναμε 3 ή 4 δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση του κεφαλαιακού κόστους όσον αφορά τις τράπεζες που θα συμμετείχαν σε αυτά τα σχέδια να, καλύψουμε τις ανάγκες. Δεύτερον, στη μελέτη επιπτώσεών σας, στη μελέτη επιπτώσεών σας αναφέρεται και πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό που κάνετε, ότι 70% των αναγκών επενδύσεων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εξυγχρονισμού των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας θα επενδυθούν. Εκπλήσωμε, τα κριτήρια έχουν έτσι, ώστε τα περισσότερα χρήματα θα πάνε για το φυσικό αέριο. Διότι, πολύ απλά, το φυσικό αέριο και αυτό σε συνδυασμό με τα 80% συγχρηματοδότησης. Και ερώτηση, όταν θα έχουμε 4 5 δισεκατομμύρια στον Ναμπούκο και τα θάψουμε στον Ναμπούκο, τα ενταφιάσουμε εκεί, θα έχουμε ψίχουλα για άλλες επενδύσεις. Και το τελευταίο, CCS, Έχουμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο επενδύσει για συγκυριακά προγράμματα και σχέδια για το CCS. Αυτό βρίσκεται στους λογαριασμούς μεγάλων επιχειρήσεων. Λίγα πράγματα έγιναν ή πολύ λίγα. Και τώρα και άλλα χρήματα θα διατεθούν. Πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση, μια εκτίμηση. Τι έγινε με εκείνο το δισεκατομμύριο που μέχρι σήμερα εμβάσαμε, δώσαμε σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο.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 και πάλι, θα ήθελα να πω, πολλά υπόσχεται αυτή η εισήγηση. Έχω κάποιες εξειδικευμένες ερωτήσεις για την αναλογία. 140 δισεκατομμύρια για ευφυή δίκτυα, για λεωφόρους, ε, λεωφόρους ενεργειακές, άλλα δισεκατομμύρια για τις υποδομές. Από πού προέρχεται αυτή η αναλογία. Τι σημαίνει αυτό για την χρηματοδότηση, ότι οι εγγυήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι με αυτή την αναλογία τροπολογία 2 προς 1 θα λειτουργήσουν 140 δις, 70 δις, 1, 2 ε, ε, προς 1. Είναι ανοιχτό αυτό το ερώτημα, δεν έχει απαντηθεί. Γιατί επιλεγμένες τέτοιες επενδύσεις θα ε, προωθούνται με αυτή την ταχεία διαδικασία και γιατί όχι όλες οι διεργασίες. Μετά ο χρόνος ε, που, κρατάνε, διαρκούν αυτά τα προγράμματα. Είναι μια διοργανωτική θα έλεγα ανομαλία μετά το South Stream. Το Ναμπούκο θα είναι δύο φορές μικρότερο από εκείνο το οποίο είχε σχεδιαστεί. Θα είναι Ναμπουκίνο, μικρός Ναμπούκο, ε, μικρός Ναβουχοδονόσορας και όχι πραγματικά μεγάλος Ναμπούκο, Ναβουχοδονόσορας. Σκεφτείτε το αυτό Επίτροπε. Με αυτό το μέσο ουσιαστικά η αρχική κλίμακα των επενδύσεων διασφαλίζεται ή όχι. Μπομπίνσκα παρακαλώ. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πίτροπε, είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο αυτό που τον εξευρωπαϊσμό της ενεργειακής μας στρατηγικής ε, θέλει να τον επιταχύνει. Εργάζομαι στην Επιτροπή Περιφερειακής συγγνώμη, στην Επιτροπή Ήτρε και θα ήθελα γι' αυτό να μου πείτε το εξής. Τι συμβαίνει τα χρήματα τα οποία έχουν εξευρεθεί για αυτό το πολύ σημαντικό σχέδιο θα δαπανηθούν εις βάρος των διαρθρωτικών κονδυλίων που τώρα θα έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη. κατάλαβα ότι ένα μέρος των κονδυλίων θα αντληθεί από εκεί, αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτών των σχεδίων, των προγραμμάτων θα πρέπει να δούμε ότι σημειώνεται έλλειψη, μείωση των κονδυλίων λόγω της άντλησης σε σχέση με τα περιφερειακά κονδύλια. Κυρία Τικάου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, Πρόεδρε, καταρχάς να σας συγχαρώ κύριε Επίτροπε μάλλον, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Έχετε ένα όραμα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε λίγο περισσότερο παρακαλώ ότι έχει σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα. Ξέρετε ότι η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι πολύτιμη για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αναφέρομαι μόνο στον Αμπούκο εδώ, υπάρχουν και άλλα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ε, δεύτερη ερώτηση. Ποιος θα διαχειριστεί το ταμείο αυτό για τις υποδομές. Θα υπάρξει κάποια νέα υπηρεσία, κάποια υπάρχουσα υπηρεσία και πώς θα συνδεθεί το ταμείο αυτό με τη διαχείριση των περιφερειακών ταμείων. Τώρα, για την ενεργειακή ένδυα, την ενεργειακή φτώχεια, πώς θα μπορέσετε να πάρετε μέτρα έτσι ώστε η ενέργεια να είναι διαθέσιμη σε μια τιμή η οποία να είναι προσιτή για τον πολίτη. Κάρινς παρακαλώ, συνάδελφε Κάρινς. σε ευχαριστώ πρόεδρε. Παρακολουθούσα τη διερμηνία η οποία είχε βραδύτερο ρυθμό από ότι ο λόγο τη ομιλήτρια που είχε ολοκληρωθεί πιο πριν. Θέλω να ευχαριστήσω, Επίτροπε. Εδώ και χρόνια κάνουμε λόγο για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Και φυσικά χωρίς ε, λειτουργούσα υποδομή, λειτουργούσες υποδομές, πράγμα που αφορά όλα τα κράτη-μέλη συνολικά και που θα συνδέει όλα τα κράτη-μέλη, δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Τώρα επιτέλους, όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει κάποιες προτάσεις. Προτάσεις, τα χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ε, για υποδομές, όχι μόνο για επιμέρους χώρες, και για τις ενεργειακές τους υποδομές μέσα σε αυτές τις χώρες θα χρησιμοποιηθούν αλλά και για την διασύνδεσή τους με τον ενεργειακό τομέα παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Κατά τούτο αυτά είναι πολύ σημαντικά για την Ευρώπη, σίγουρα. Έχω όμως μια ερώτηση. Ποια αναλογία είναι εκείνη που βλέπετε εσείς ή πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ισχύσει για τα προγράμματα και σχέδια στην ίδια την Ευρώπη και για προγράμματα όπως το Ναμπούκο εκτός Ευρώπης. Ποια θα είναι η αναλογία ή μήπως αυτό το, τα 9 δισεκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Κυρία Ποδηματά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε. Ε, θέλω και εγώ από την πλευρά μου να υπογραμμίσω ότι θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την πρωτοβουλία αυτή για το πακέτο των ε, ενεργειακών υποδομών και για την προώθηση των στόχων της Ένωσης για την ε, ενέργεια και το κλίμα και για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Θα προσέθετα και για την υπέρβαση της σημερινής κρίσης και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας διότι κύριε επίτροπε δεν θεωρώ τυχαίο ότι η προώθηση ενεργειακών σχεδίων ε, περιλαμβάνεται στον οδικό χάρτη που παρουσίασε ο πρόεδρος της επιτροπής την περασμένη τετάρτη για την έξοδο της ε, ε, ευρωπαϊκής ένωσης και της ευρωζώνης από την κρίση και την δρομολόγηση μιας πορείας ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. ένα από τα πιο κέρια ζητήματα είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης επισημάνθηκε από πολλούς συναδέλφους Είπατε εσείς στην παρουσίασή σας ότι το κόστος και οι κίνδυνοι πρέπει να σταθεροποιηθούν με ε, ευρωπαϊκή ρύθμιση και ήθελα να σας ζητήσω αν μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Με δεδομένο ότι στην παρούσα συγκυρία ε, η χρηματοδότηση δεν είναι εύκολο να προωθηθεί ούτε μέσω προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων λόγω περικοπών ε, αλλά ούτε και από τον ιδιωτικό τομέα διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά παράπονα σε πολλές χώρες ε, ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν διοχετεύει επαρκή ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και ειδικότερα ε, σε προγράμματα και σχέδια σαν αυτά που συζητάμε. Δεδομένου ότι γίνεται μια συζήτηση για την ενίσχυση των τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συζητάμε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση σε αυτή τη φάση θα σκέφτεστε ε, να ε, υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να θεσπιστούν κάποιες προτεραιότητες, κάποιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών τραπεζών ώστε να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα έργα περιλαμβανομένων αυτών που συζητάμε σήμερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεύτερο, ολοκληρώνω κύριε ε, Πρόεδρε, Υπάρχουν σκέψεις για μεγάλα έργα ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη, ειδικά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γνωρίζετε για το σχέδιο δημιουργίας μεγάλων ηλιακών εγκαταστάσεων στον Ευρωπαϊκό Νότο, στην Ελλάδα, για εξαγωγή ηλιακής ενέργειας στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Υπάρχουν τρόποι η Επιτροπή να ενθαρρύνει και να προωθήσει αυτού ναι. του είδους πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον Επίτροπο ότι επιτέλους έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και κάποιες πράξεις στο συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε βαρεθεί τα λόγια μέχρι τώρα. Αυτά τα προγράμματα, αυτά τα σχέδια είναι νομίζω ουσιαστικά, αντικειμενικά έχουν σχεδιαστεί και είναι και εφικτά. Υπάρχει ένα θέμα σχετικά με τη χρηματοδότησή τους, αλλά νομίζω ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμφέρον για να προχωρήσει η κατάσταση. Όταν μιλάμε βέβαια για ενιαία αγορά στον τομέα της ενέργειας, νομίζω ότι κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει ενιαία αγορά. Αν δει κανεί τις ανατολικές χώρες, αν δει κανεί τις χώρες της Βαλτικής, ε, είναι προφανές ότι είναι απόλυτα εξαρτημένες από μία συγκεκριμένη πηγή προμήθειας φυσικού αερίου. Συνεπώς δεν υπάρχει πραγματική ενιαία αγορά και μάλιστα σε κάποιες περιοχές εφόσον θέλουμε να διασφαλίσουμε την προμήθεια ενέργειας η συμμετοχή κοινοτική μπορεί να χρειαστεί να φτάσει μέχρι και το 80%. Επιμένω στην περιοχή της Βαλτικής εκατομμύρια κυβικών μέτρων φυσικού αερίου είναι απαραίτητα για να συνεχιστεί κανονικά η δραστηριότητα η οικονομική στην περιοχή. Σώσα Βάγνερ παρακαλώ. Γράφειες. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Για να επιμείνω και να εμείνω σε κάτι που αναφέρθηκε πολλές φορές εδώ που είναι το πρόβλημα των διαδικασιών αδειοδότησης στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι ο στόχος του εγγράφου που υποβάλλει η Επιτροπή είναι καλός. Διαρωτώ με, αυτές οι προθέσεις θα αντιστοιχούν με την δράση από πλευράς των κρατών και με τις δυσκολίες που δημιουργούν η εσωτερική νομοθεσία στα κράτη-μέλη ιδιαίτερα με αποκεντρωμένες χώρες, με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό αποκέντρωσης. Ένα άλλο θέμα, Επίτροπε, είναι το θέμα της αντίθεσης των πληθυσμών, του λαού σε σχέση με τέτοια προγράμματα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επιμείνουμε πολύ, επειδή μπορούν να οδηγήσουν να αποτύχουν όλε οι καλέ προθέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλε οι καλέ προθέσει που έχουμε όλοι. Ακριβώ σαν συνέπεια της αντίστασης και αντίδρασης που οργανωμένοι πολίτες ασκούν σε σχέση με αυτά τα μεγάλα προγράμματα και σχέδια. Και τελευταίο θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου, να εκφράσω τη θλίψη μου δημόσια ότι η Βυρική Χερσόνησος έχει εξαφανιστεί από το έγγραφο που έχει παρουσιαστεί. Ελπίζω ότι θα επανέλθει, θα ξανάρθει και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη θέση της όπως της αξίζει. Ευχαριστώ. Herzog παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά ιδιαίτερα τον κύριο Επίτροπο που παρίσταται εδώ σήμερα. Πολλές ερωτήσεις θα είχα, όμως οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν ήδη διατυπώσει τις περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις και γι' αυτό θα ήθελα να επικεντρωθώ σε εκείνα τα σχέδια και προγράμματα που είναι διασυνοριακά και αφορούν περισσότερες χώρες που διασυνδέονται μέσω αυτών. Με τι μπορούμε να υπολογίζουμε όσον αφορά τις διάφορες συμβάσεις Ποιος είναι εκείνος που θα είναι υπεύθυνος για αυτές τις συμβάσεις τελικά. Και τίθεται το ερώτημα, είναι ρεαλιστικό να αναμένει κανείς ότι τέτοιες συμβάσεις και συμβόλαια θα συναφθούν στο μέλλον περαιτέρω για τέτοιου είδους μεγάλα σχέδια και προγράμματα. Είδαμε πόσο δύσκολο ήταν για παράδειγμα υπό το πλαίσιο της Euronest να ξεκινήσει μια τέτοια διεργασία. Ευχαριστώ. Καρβάλιο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο Πράγματι το θέμα αυτό έπρεπε να το συζητήσουμε. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω επίσης γιατί θέτει και τον διάδρομο βορρά-νότου στην ημερήσια διάταξη. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για τον νότο της Ευρώπης αλλά και συνολικά για την Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας λίγο και στην Ιβυρική Χερσόνησο. Αναφερθήκατε επίσης και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Υπάρχουν πολλοί τερματικοί σταθμοί, οι οποίοι όμως δεν είναι επαρκείς. Παρ' όλα αυτά, στην Ιβερική Χερσόνησο έχουμε 7 τέτοιους τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου υγροποιημένου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάλλιστα και για την υπόλοιπη Ευρώπη με τις σωστές διασυνδέσεις. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω με την, την σημασία που έχει η αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας ε, ποσοτήτων φυσικού αερίου και καυσίμων γενικότερα. Βίνκλα. Ευχαριστώ ε, και σας κύριε Πρόεδρε και τον κύριο Επίτροπο για τις ρεαλιστικές προτάσεις. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα <clears throat> η διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και εγκρίσεως. Μάλλον τα γνωρίζετε αυτά που θα πω, αλλά στην επανένωση των δύο Γερμανιών, να το πω έτσι απλά, είχαμε σημαντικές εμπειρίες από την διασύνδεση των οδικών δικτύων που μέσα σε λίγο χρόνο επέτρεψε η υποδομή στην Γερμανία παρόλο που ήταν πάρα πολύ διαφορετικά τα συστήματα και να λειτουργήσει αλλά και να χρηματοδοτηθεί. Ίσως εν μέρη αυτό μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για το δικό σας Connecting Europe στον τομέα της ενέργειας. Μάλιστα, θα δώσω πάλι τον λόγο στον Επίτροπο και με την παράκληση να απαντήσει βέβαια σε σύντομο χρόνο. Στις χώρες μέλη ξεκινούμε από πολύ διαφορετικές προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την συνταγματική, τη συνταγματική κατοχήρωση της ιδιοκτησίας γης καθώς και τις διάφορες δικαστικές δικαιοδοσίες. Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι στην Μάλτα οι επιμέρους ειδικέ αρχές και οι δικαστικές αρχές είναι στον ίδιο αριθμό όπως στη Γαλλία. Σε ορισμένες εθνικές συνταγματικές τάξεις έχουμε ξεκάθαρους κανόνες που επιβάλλουν και δικαιώματα αλλά και υποχρώσεις στην ιδιοκτησία. Έτσι, η διαδικασία των τριών ετών δεν μπορεί να εφαρμοστεί, να ρυθμιστεί δηλαδή σχηματικά πανευρωπαϊκά με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να θέσουμε το πλαίσιο των τριών ετών και η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια του εθνικού εκάστοτε συνταγματικού δικαίου καθώς και των υπολείπων νόμων και θα πρέπει να μας εξηγήσουν οι χώρες μέλη με ποιον τρόπο θα τηρήσουν το πλαίσιο των τριών ετών. Ασφαλώς θα χρειαστεί ενίσχυση του ειδικού προσωπικού, των οργανογραμμάτων δηλαδή των ειδικών ε, αρχών θα χρειαστεί και ίδρυση ειδικών τμήματων των δικαστηρίων για την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. Εμείς περιοριστήκαμε σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση στην διαμεθοριακή υποδομή. Γιατί? Διότι εκεί πρόκειται για ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Σε καμία χώρα μέλος δεν απαγορεύεται, αντιθέτως με το μοντέλο που προωθούμε, που υποτίθεται ότι θα είναι ένα πρότυπο, θα έχει κάθε χώρα μέλος την δυνατότητα να προβλέπει την επιτάχυνση αυτή για σημαντικά έργα υποδομής τα οποία σχεδιάζονται μέσα στην επικράτειά του. Καθώς επίσης και για δικτύα διανομής. Μιλούμε τώρα για τις διασυνδέσεις, αλλά υπάρχουν και της ίδιας σημασίας τα εθνικά δίκτυα διανομής. Εκεί μοναδικός αρμόδιος είναι ο εθνικός νομοθέτης, ο οποίος μπορεί να προβλέψει και πρέπει να προβλέψει διαδικασίες επιτάχυνσης. Κύριε Τούρμες, για τα 9 δισεκατομμύρια, 8 συν 1, είμαι απολύτως ανοιχτός. Το 1 δισεκατομμύριο με το οποίο θέλουμε να ε, χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για να ε, δώσει, να, να δώσει την ευκαιρία να υπάρξουν και άλλες χρηματοδοτήσεις. Άλλωστε ασκείται και σημαντική κριτική. Γι' αυτό Θέλουμε να αρχίσουμε μια προσπάθεια μαζί με τις τράπεζες εταίρους και αν αποδειχθεί η αξία του μοντέλου αυτού θα την εφαρμόσουμε με ετήσιες δόσεις. Ετησίως. Λέω λοιπόν ήδη σαφώς ότι μετά από ένα-δύο χρόνια εφόσον αποδειχθεί ότι λειτουργεί θα αυξήσουμε τα χορηγούμενα κονδύλια και θα μειώσουμε αντιστοίχως εφόσον έχουν τα ποσά αυτά απολεστεί. Ναμπούκο δεν θίγεται από τα σχέδια αυτά. Ο Ναμπούκο θα υλοποιηθεί με το EPPA. Και το ίδιο για το, για τον νότιο διάδρομο. Θα πρέπει στους επόμενους μήνες να έχουμε απόφαση. Όχι όμως πλέον για την περίοδο 2014-2020. Και για τα CCS, τα, το συζητήσουμε τον Νοέμβριο, θα σας υποβάλουμε τον ενδιάμεσο απολογισμό. Εκεί έχουμε προβλέψει μόνο εντός εισαγωγικών 2-2,5 δις, 140 περίπου ε, ε ρεύμα, 70 για το αέριο. Τα κονδύλια αυτά, ένα δισεκατομμύρια που μας δώσατε για 6-7 έργα της, δική δικής μου ευθύνης, αλλά για, το, για, την για τον επιτόπο Hildegard Από αυτά πληρώνονται μόνο σύμβουλοι. Δεν μπαίνουν σε τράπεζες, δεν αποδίδουν τόκους. Είναι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θα πληρώνονται καταδόσεις ανάλογα με την πρόοδο του έργου στα ε, έργα επίδειξης δηλαδή, όπου ορισμένα προχωρούν καλά και άλλα βρίσκονται ακόμη στην φάση του σχεδιασμού. Τα 140 για το ηλεκτρικό και 70 για το φυσικό ε, αέριο δεν είναι η δεσμευτικά όσον αφορά τα 9 δις από πλευράς μας. Μπορεί για το φυσικό αέριο και για πύργους φυσικού αερίου να δαπανηθούν περισσότερο από το 1 τρίτο στο τέλος τέλος πάνω από τρία δις. Αλλά αυτό εξαρτάται τελικά από τους καταλόγους προτεραιοτήτων πρώτων. Δεύτερον, και κατά πόσον σε ποιο βαθμό αυτά τα προγράμματα για να είναι ικανά να τύχουν δανειοδότηση από τράπεζε θα χρειάζονται και συγχρηματοδότηση από εμά. διασυνδέσεις ε, όσον αφορά τα αστικά κέντρα Ρότερνταμ, Άμστερνταμ προς Ντόρτμουντ. Ε, Διασύνδεση δηλαδή, α το πω έτσι, των κάτω χωρών και της γερμανίας. Κάθε διασύνδεση είτε είναι ηλεκτρική ενέργεια είτε φυσικού αερίου δεν θα χρειάζεται ούτε ένα ευρώ διότι μεταξύ των δύο αυτών μετροπόλεων υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες που από πλευρά τη ίδια τη συμμετοχή στην αγορά θα έχουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Και έχουμε και άλλα προγράμματα κοινού συμφέροντος που χρειάζονται κατεπηγόντως 10 έως 80% υποστήριξη, συγχρηματοδότηση εδώ όλα θα εξαρτώνται πάντα από το τι θα μπορούν να υπομισθούν οι καταναλωτές. Τι μπορεί κανείς μέσω υψηλότερων τιμών για το ηλεκτρικό και το φυσικό αέριο να καλυφθεί και κατεπηγόντως πρέπει να αποφύγουμε να μην εκραγούν οι τιμές προς τα πάνω του ηλεκτρικού και της, ε, του φυσικού αερίου. Και φυσικά εδώ έχουμε στην πρόταση για τον προϋπολογισμό ε, την αντιδιαστολή προς οποιαδήποτε άλλη δαπάνη. Έτσι τίθεται το αν τα 40 δις και μέσα σε αυτά τα 40 δις θα έχουμε 10 δις για την ενέργεια από το διαρθρωτικό πακέτο μέτρων. Και ναι και όχι. Θα μπορούσε και κάποιος πολιτικός για τη γεωργία να πει στον πρώτο ή δεύτερο πυλώνα στην ΚΑΠ μας λείπουν χρήματα. Όμως αυτό είναι το υψηλότερο έργο συντονισμού των δημοσιονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό πάλι συναρτάται με το θέμα του πόσο μεγάλο θα είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1,0% του ΑΕΠ, 1,05% του ΑΕΠ. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι αυτό το ποσοστό. Θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι σήμερα. Θα είναι το ίδιο το ποσοστό όπως σήμερα ή κιόλα και μικρότερο. Και γι' αυτό προτεραιότητες στη δημοσιονομική πολιτική πρέπει να τεθούν όπου πιστεύουμε ότι για την ενέργεια δέκα δις πρέπει να διατεθούν διότι η ενέργεια είναι σημαντικό θεμέλιο για την προστασία του περιβάλλοντος, την διασφάλιση της ευημερία μας και πουθενά αλλού δεν έχουμε τόσο μεγάλες ανάγκες όσο στον τομέα των υποδομών για την ενέργεια. Έτσι λοιπόν οι υποδομές για τις μεταφορές παρότι υποστηρίζουμε το δικό δίκτυο και τους σιδηροδρόμους περαιτέρω στην Ευρώπη σε σχέση με το ηλεκτρικό και το φυσικό αέριο. Εδώ έχουμε ιστορικό καθήκον να καλύψουμε τα κενά και τις ανάγκες. Ερωτήθηκε ποια προγράμματα ακόμα στα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Θέλουμε συνειδητά στις μεγάλες αυτές περιφέρειες και η Ισπανία, Γαλλία, η Ισπανία, Πορτογαλία ως μεγαλύτερες περιφέρειες και γιατί όχι η Ισπανία, Μαρόκο και θέλουμε τα κράτη-μέλη σε σχέση με τους παρόχους των δικτύων και των ε, ενεργειακών ε, μονάδων παραγωγών να συμμετάσχουν. Σας λέω, αν είχαμε έναν ολοκληρωμένο κομμένο και ραμμένο κατάλογο προτεραιοτήτων, τα κράτη-μέλη και κάποιοι ευρωβουλευτές μόνο θα έλεγχαν ποια κονδύλια θα διατεθούν ανά χώρα. Τελεία και παύλα. Και τι θα γινόταν αν είχαμε λιγότερα από ό,τι εκείνα τα οποία θα χρειαζόντουσαν τότε η πρότασή μας ουσιαστικά εκ προημίου θα υπονομευόταν, θα καταστρεφόταν. Πρέπει να είμαστε συνετοί. Ας πάρουμε τη χώρα μου, τη Γερμανία. Η Γερμανία, από ό,τι γνωρίζω εγώ, είναι βέβαιο ότι στον ενεργειακό τομέα για τις υποδομές, για την συγχρηματοδότηση θα ανακτήσει λιγότερα κονδύλια από ό,τι θα πληρώσει γενικά. Γιατί, διότι μια χώρα στον πυρήνα, στην καρδιά της Ευρώπης, με μεγάλο αριθμό πληθυσμού, με βιομηχανία, με μεγάλα δίκτυα υποδομών που πρέπει να ε, χρηματοδοτηθούν και για τις τιμές των προϊόντων που θα μεταφέρονται που πρέπει να είναι προσιτές. Αντίστροφα όμως, οι βαλτικές χώρες, η Μάλτα, και η Ελλάδα αντίστροφα δεν θα μπορέσουν να, να πετύχουν την ολοκλήρωσή τους και την ένταξή τους χωρίς συγχρηματοδότηση. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα συνετά και ε, με πρόβλεψη ότι από τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιταλία επιχειρήσεις όπου συνεργάζονται και δρούν στην ενεργειακή αγορά και συμμετέχουν σε αυτήν η ένταξη των αγορών αυτών και στην ε, πολιτική, τη βιομηχανική πρέπει να εξεταστεί. Καλείται εδώ ε, να εκφραστεί με ευφυή τρόπο η δράση μας και η αλληλεγγύη μας. Και το ερώτημά σας ως τελευταίο σημείο σήμερα τις ε, περαιτέρω ερωτήσεις τις, την επόμενη, τις επόμενες εβδομάδες ε, θα τις ε, απαντήσω. Αν θα έχουμε τα κονδύλια για την Ευρώπη των 27 κρατών μελών ή θα αφορούν και τις τρίτες χώρες. Αυτό το επίκεντρο θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα αλλά το να επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο στην ευρωπαϊκή επικράτεια θα ήταν λάθο. Παράδειγμα, αν τώρα με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια θέλουμε να είμαστε σοβαροί με του στόχου μα στην Ελλάδα και με το Task Force, είχα και συζήτηση με τον κύριο Ράιχενμπαχ και έχουμε την πρόταση οι ανανεώσιμε πηγέ και στην υποδομή για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια να προαχθούν και αυτό θα αποτελεί και μέρος του, του σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων, τότε πρέπει ταχύτερα σε σχέση με την αγορά να προβλέψουμε δίκτυα προς και από την Βουλγαρία, Ρουμανία, Αυστρία, Γερμανία και να ολοκληρώσουμε αυτές τις διασύνδεσεις. Καλό θα ήταν για τις αγορές μας, για την Ελλάδα ιδιαίτερα, την επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια να την προβλέψουμε και να την συγχρηματοδοτήσουμε. Και στη Σερβία και Μαυροβούνιο όταν θα βρίσκονται εκεί τέτοιες διασυνδέσεις υποδομών που δεν είναι ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σίγουρα τα επόμενα δέκα χρόνια θα μπορούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό και αυτά τα δίκτυα θα μπορούν με μια συγχρηματοδότηση να ολοκληρώνουν το ηλεκτρικό δίκτυο μεταξύ Ελλάδας, Σλοβενίας, Δυτικών Βαλκανίων εργαλείων. Ή ένα άλλο παράδειγμα. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί με τις προθέσεις μας για την εταιρική σχέση στα ενεργειακά με, το νότια, με τη Νότια Μεσόγειο, τότε <clears throat> μέσω καλωδίων, μέσω της Μεσογείου προς την Ισία, από την Τινησία Αλγερία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να πούμε ότι τέτοια καλωδίωση θα είναι προς όφελός μας και μια τέτοια συγχρηματοδότηση παρότι βρίσκεται εκτός των κρατών μελών είναι προς ευρωπαϊκό όφελος και πρέπει να ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση και συνεισφορά σας και είμαι στη διάθεσή σας να εμβαθύνουμε σε οποιαδήποτε πτυχή αυτών των θεμάτων στο μέλλον. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος όλων θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά κύριε Επίτροπε για αυτές τις πρώτες πληροφορίες. Κυρίως επειδή και γοργά ε, είχαμε τις ε, προτάσεις αυτές και θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο με ζήλο στο μέλλον. Επόμενο σημείο. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη Διασύνδεση και έχουμε ήδη συζητήσει διάφορα πράγματα γι' αυτό και σήμερα για άλλη μια φορά έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες. Ο κύριος Τσίτσεστερ σήμερα παρακολύεται, δεν μπορεί να παραστεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν αλλάξαμε τα θέματα στην ημερήσια διάταξη επειδή έγκαιρα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Επιτρέψτε μου να επισημάνω και κάτι άλλο. Έχουμε μία ομάδα αρκετών θεμάτων που τίθενται. Την τελευταία φορά τα είχε παρουσιάσει ο κύριος Τσίτσεστερ. 200 τόσες τροπολογίες. Είναι σαφές και το χρονοδιάγραμμα. 10 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε προς έγκριση. Να ρωτήσω τους χειώδεις εισηγητές. Αν τα βλέπω καλά ο συνάδελφος Έλερ θα αναλάβει τα θέματα της παρουσίασης του κυρίου Τσίτσεστερ. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο τώρα. Παρακαλώ, είναι δυνατόν να υπάρξει ησυχία στην αίθουσα. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι πρέπει να φλιαρούν όταν βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Δεν μπορείτε να βγείτε έξω αν θέλετε να συζητήσετε. Είναι μια ερώ... ένα θέμα ευγένειας και φιλικής αντιμετώπισης των συναδέλφων. Ο κύριος Έλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, δεν μπορώ ακριβώς να πάρω τη θέση του εισηγητή, αλλά μιας και ο κύριος Τσίτσεστερ δεν μπορεί να είναι ανάμεσά μας σήμερα, θα προσπαθήσω να ξεκινήσω μια πρώτη συζήτηση για τις τροπολογίες από πλευράς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ίσως, αλλά και λίγο γενικά. Στην ουσία όλοι πλέον μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ενισχύσει το θέμα της κυβερνοασφαλείας. Θέλει να ενισχύσει το ρόλο της αρμόδιας υπηρεσίας, η ΕΝΙΣΑ, οι αρχές της ΕΝΙΣΑ ήταν μια θα έλεγα μορφή συμβιβασμού ανάμεσα σε ορισμένες χώρες οι οποίες δεν ήταν σίγουρες για το ρόλο της ΕΝΙΣΑ και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες είχαν συγκεκριμένες απόψεις και ενδιαφέροντα. Νομίζω όμως ότι η ΕΝΙΣΑ απέδειξε ήδη ότι αξίζει τον κόπο και αξίζει τον κόπο να ενισχυθεί. Η κατάσταση είναι πολύ πιο δραματική θα έλεγα από ότι όταν είχαμε πει ξεκινώντας τη συζήτηση. Αν δει κανεί τον αριθμό των τροπολογιών θα διαπιστώσει ότι μπορεί να τις κατατάξει σε τρία διαφορετικά κεφάλαια. Πρώτον υπάρχουν οι τροπολογίες οι σχετικές με την εντολή της ενίσα και τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θέλουμε να διευρύνουμε την εντολή. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για μια υπηρεσία με εκτελεστική εντολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, πάντα τα κράτη-μέλη θα είναι αρμόδια. Αλλά παρόλα αυτά εμείς θέλουμε να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες και την αποτελεσματικότητα και τις προοπτικές της ενίσα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Καταρχάς θεωρούμε ότι η ΕΝΙΣΑ δεν έχει μία αποκλειστικά εντολή. Το θέμα δεν είναι μόνο η σχέση της ΕΝΙΣΑ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία τίθενται. Αλλά έχουμε να κάνουμε με μία κατάσταση μερικές φορές η οποία θα έλεγα ξεπερνάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν κάποιες χώρες θέλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με την ΕΝΙΣΑ και να ζητήσουν την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΝΙΣΑ, τότε πρέπει να έλθει αρρωγός τους και το θέμα δεν είναι εδώ η τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΝΙΣΑ και τα υπόλοιπα όργανα και τις εξωτερικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει η ΕΝΙΣΑ να προσπαθήσει να διαμορφώσει σωστά τα προγράμματα ασφαλείας και στον τομέα των τηλεπληροφοριών και στον τομέα της πληροφορικής δεν συμμετέχει καν στις υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή ελέγχουν το θέμα της ασφαλείας στον κλάδο της πληροφορικής. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν έχει λογική. Θέλουμε λοιπόν εμείς μέσα από τις τροπολογίες να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για εκτελεστικό όργανο, για εκτελεστική υπηρεσία, παρόλα αυτά πρέπει να την ενισχύσουμε, να διευρύνουμε τις αρμοδιότητές της και να διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητά της με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα θα έλεγα. Η δεύτερη ομάδα των τροπολογιών αφορά την διάρκεια την χρονική της εντολής. Εδώ υπάρχουν εντελώς διαφορετικές θέσεις. Κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται για μία μόνιμη εντολή προς μία εξωτερική υπηρεσία πλέον. Αυτό δεν είναι κάτι το καινοφανές, αλλά είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να επικυρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η διάρκεια της εντολής κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται και εξαρτάται από το θέμα ε, με το οποίο ασχολείται η συγκεκριμένη υπηρεσία. Λοιπόν, μια συμβιβαστική πρόταση στον τομέα αυτό είναι να διευκρινίσουμε ότι εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι το θέμα της ε, ασφάλειας στον τομέα του κυβερνοχώρου είναι ένα θέμα μακροπρόθεσμου και πρέπει να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη χρονική προοπτική. Συνεπώς Είτε μπορούμε εμείς να δεχθούμε την απεριόριστη χρονικά εντολή, αλλά με μια ρήτρα αναθεώρησης ή επικαιροποίησης αναπενταετία, συγγνώμη, ή να αποφασίσουμε για μια χρονική περίοδο δεδομένη και μετά να αποφασίσουμε πια τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα όταν ε, λήξει η περίοδος αυτή. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το θέμα αυτό άπτεται αν θέλετε ε, της οργανωτικής μορφής την οποία θα πάρει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Η φύση θα έλεγα της ε, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι κάτι το οποίο είναι σαν κινούμενη άμμος. Αλλάζει συνεχώς σχήμα, αλλάζει συνεχώς μορφή. Η δομή λοιπόν της ενίσας στην παρούσα φάση θα πρέπει να ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο τις αρχές της προστασίας αυτής της, του κυβερνοχώρου γενικότερα. Δεν ξέρω τι δομές και τι σχέσεις θα διαμορφωθούν στο μέλλον. Σαν παράδειγμα μπορεί να υπάρξουν δομές στο ΝΑΤΟ που να ασχολούνται με το συγκεκριμένο αυτό χώρο. Ίσως λοιπόν τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 5-6 χρόνια, να αποφασίσουμε ότι απαιτείται μια νέα δομή, μια ευρύτερη δομή, μια πιο αποτελεσματική δομή. Ξέρετε τι συνέβη στις Ηνωμένε Πολιτείες. Μέσα σε μια πενταετή περίοδο οικοδόμησαν την δική τους, αν θέλετε, αρχιτεκτονική για την προστασία του κυβερνοχώρου. Χρειάστηκε λοιπόν κάποιος χρόνος. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε στην αρχή μιας τέτοιας χρονικής περίοδου σε αυτή τη φάση. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τι μορφή θα πάρουν οι μελλοντικές εξελίξεις και αν δούμε ότι κάτι τέτοιο ε, είναι εφικτό μπορούμε να χορηγήσουμε μία περίοδο εντολής χωρίς όρια. Από την άλλη, αν δούμε ότι είναι δύσκολο να διαμορφώσουμε μια συγκεκριμένη εικόνα, τότε ας δώσουμε μια προθεσμία συγκεκριμένη και από εκεί και πέρα θα δούμε. Το τρίτο θέμα, η τρίτη ομάδα των τροπολογιών. Εδώ είμαι απογοητευμένος από τις διαπραγματεύσεις the με την ελληνική κυβέρνηση. Όλος αυτός ο αγώνας για την έδρα της Ενίσα δεν έπρεπε να υπάρξει. Υπήρξε μια συμβιβαστική πρόταση η οποία προτάθηκε ανάμεσα σε διάφορα κράτη-μέλη το θέμα δεν είναι πού ε, είναι η έδρα της συγκεκριμένη υπηρεσία. Το θέμα είναι η λειτουργικότητα της υπηρεσίας αυτής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμβιβαστική λύση αποδεκτή από όλους τους εμπλεκομένους. Ίσως τελικά μπορεί να παραμείνει η ενίσα στην Κρήτη με κάποιο πως πιο μόνιμο και διοικητικό προσωπικό, να υπάρχει ένας κλάδος στην Αθήνα με το λειτουργικό κομμάτι, γιατί πρέπει να ταξιδεύουν συχνά, πρέπει να μετακινούνται συνεχώς. Θυμίζω ότι η ενίσα δεν είναι να κάθεται κάποιος μπροστά στη, στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτό είναι κάτι που το κάνουν και τα κρατημέλη μόνα τους. Η ΕΝΙΣΑ είναι μια υπηρεσία η οποία προσπαθεί να σταθμίσει τα συμφέροντα. Είναι μια πλατφόρμα συνδυασμού αν θέλετε ενδιαφερόντων. Και ιδιαίτερα αν θέλουμε να διευρύνουμε την εντολή της ΕΝΙΘΑ τότε είναι απαραίτητο η υπηρεσία αυτή να είναι λειτουργική. Λοιπόν, ας παραμείνουμε λοιπόν εκεί που είμαστε. Ας υπάρξει μια αντένα λειτουργική ισχυρή στην Αθήνα και ένα γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες. Αλλά αυτή η συζήτηση είναι λίγο περιττή. Εμείς εμένουμε για πολιτικούς συμβολικούς ε, λόγους σε κάποιες απόλυτες θέσεις λέγοντας ότι όλα θα πρέπει να είναι στην Κρήτη, όλα θα πρέπει να γίνουν στην Κρήτη. Αυτό δεν είναι συμβιβασμός. Το θέμα είναι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι πλήρως λειτουργικό. Εγώ ήρθα μόλις χθες από τη Ουάσιγκτον, σήμερα το πρωί έφτασα από τη Ουάσιγκτον. Ε, οι διαπραγματεύσεις με το Πεντάγωνο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας στον τομέα της πληροφορικής με τους Αμερικανούς και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ε, η ΕΝΙΣΑ ως λειτουργεί σήμερα δεν είναι πλήρως λειτουργική. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο για τους ανθρώπους της να πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο. Το θέμα είναι να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική θέση. Να μην κολλάμε σε συμβολικές παραστάσεις Πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά. Πρέπει να σταθούμε πρακτικά απέναντι στα προβλήματα. Και αν υπάρχει παρακαλώ λίγος χώρος, λίγο περιθώριο κίνησης από πλευράς ε, της ελληνικής κυβέρνησης, θα προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε. Δεν είναι αυτό το βασικό μας πρόβλημα. Ο Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που αναγκάζομαι να σας διακόψω γιατί έχουμε στις 10 την ψηφοφορία. Κύριε Βαλιάν. Έχουμε τώρα τις συμβαστικές τροπολογίες. Λίγα λόγια, να σας πω, για την διάρκεια της ε, θητείας ε, θα υπάρχουν δύο επιλογές. Να υπάρχει όμως και έγκαιρη ε, αξιολόγηση από πλευράς Κομισιών και Κοινοβουλίου για την λειτουργία του οργανισμού για να μπορέσει να λειτουργήσει ως πλήρης, πλήρης οργανισμός της ε, Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τους ε, στόχους που θα πρέπει να ε, εξυπηρετεί η ΕΝΙΣΑ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να περιλαμβάνεται η κυβερνοασφάλεια και η προστασία δεδομένων μέσα στα πλαίσια δηλαδή των αρμοδίτων της ΕΝΙΣΑ και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβει λειτουργικές, λειτουργικά καθήκοντα. Αλλά βέβαια η διάκριση ανάμεσα σε λειτουργικά και μη, η επιχειρησιακά και μη καθήκοντα είναι πολύ λεπτή. Ήδη το 2010 έγινε η πρώτη αξιολόγηση. Με όλους τους φορείς θα πρέπει να υπάρξει ένα είδος επιχειρησιακής, επιχειρησιακού καθήκοντος. Από την άλλη μεριά δεν νομίζω να υπάρχει κίνδυνος να μπορεί δηλαδή η Ένισα να στηρίζει για την ασφάλεια των υποδομών και τα θεσμικά όργανα. Τώρα αυτό θα απαιτεί βέβαια πλήρους χρόνου όλη την εβδομάδα ε, δραστηριότητα. Τώρα για την έδρα. Νομίζω ότι δεν είναι υπόθεση του Κοινοβουλίου να υποδείξει πού θα πρέπει να είναι η έδρα της, ε, του οργανισμού αυτού. Ας αναλάβει το Συμβούλιο να ξανασυζητήσει το θέμα. Ο συμβιβασμός με το γραφείο στην Αθήνα και ε, μία αντένα στις Βρυξέλλες μου φαίνεται λογική, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο κρίσης και των οικονομικών προβλημάτων της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχω τόσο μεγάλη διάθεση να το συζητήσω, ούτε είναι σαφές για μένα αν οποιασδήποτε δεσμεύσεις ή υποσχέσεις δοθούν τώρα θα είναι αρκετές. Ας το, αρχί, ας το ξανασυζητήσει λοιπόν το Συμβούλιο και ας εκφράσουμε εμείς τις δικές μας ιδέες. Αλλά νομίζω δεν είναι δική μας υπόθεση. Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστούμε κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω εκ προημίου ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή ενίσα, με μια ισχυρή από πλευρά οργανισμού τέτοια υπηρεσία, διότι ο τομέας του δικτύου θα είναι όλο και πιο σημαντικός και σήμερα και στο μέλλον. Γι' αυτό μακροπρόθεσμα πρέπει να τα προσεγγίσουμε όλα αυτά σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Γι' αυτό εμείς μια εντολή για μια απεριόριστη περίοδο θα υποστηρίζαμε, όπου οι εργασίες, το έργο της ΕΝΙΣΑ κάθε πέντε χρόνια θα αναθεωρούνται ώστε να επικαιροποιούνται όσον αφορά την ανταπόκριση προς τις νέες προκλήσεις. Δεύτερο, εκπνοή της εντολής. Πιστεύω ότι εδώ είναι αναγκαίο η ΕΝΗΣΑ να μπορέσει λειτουργικά να έχει τις ικανότητες εκείνες να είναι σε θέση αποτελεσματικά τις δραστηριότητες των κρατών μελών όσον αφορά τα δίκτυα και την ασφάλεια των δικτύων να υποστηρίζει όλες αυτές τις δραστηριότητες και δράσεις θέλω ρητά και κατηγορηματικά να πω ότι εδώ δεν πρόκειται για συντονισμό της εργασίας στα κράτη-μέλη, υποκατάσταση των πρωτοβουλίων των κρατών μελών. Δηλαδή η ίδια η ΕΝΕΣΑ δεν θα πρέπει να υποκαθιστά άλλες, άλλους οργανισμούς των κρατών μελών για την ασφάλεια των δικτύων. Είναι αναγκαίο όμως να συνεισφέρει η ΕΝΕΣΑ για την εκπόνηση των ευρωπαϊκών εκείνων προδιαγραφών για την ασφάλεια των δικτύων γιατί μόνο έτσι μπορούμε να συνεισφέρουμε για τη διεθνή συνεργασία από πλευράς μας, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και συλλογή πληροφοριών θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πληροφορίες δηλαδή που τα κράτη-μέλη ε, τα ίδια χρησιμοποιούν και έχουν ανάγκη να διατίθενται προς, τις, ε, προς τα πανεπιστήμια, προς τους οργανισμούς και άλλους φορείς, ώστε να εξευρεθούν λύσεις, ώστε στο μέλλον τα θέματα ασφάλειας να καλύπτονται όσον αφορά την τεχνολογία ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα θέματα ασφάλειας δικτύων. Είναι αναγκαίο επίσης να μεριμνήσουμε περαιτέρω, ώστε η ΕΝΗΣΑ να είναι σε θέση τελικά πανευρωπαϊκά να μπορεί να δρά και να λειτουργεί χρειαζόμαστε ίσως ε, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ένα είδους, ε, ας το πω έτσι, θηρίδα ή ε, διαμεσολαβητή. Και πρέπει να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού θα έπρεπε να εισραίει στον τομέα της ασφάλειας δικτύων ως ε, θέμα. Λιγότερο τα κονδύλια θα πρέπει να εισραίουν προς τη διοίκηση και γι' αυτό έχω καταθέσει και κάποιες τροπολογίες για να διασφαλίσω αυτές τις πτυχές. Και δύο λόγια για, χρονοδια... για την έδρα. Η έδρα θα είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε για τα κριτήρια κάποτε για την, ε, τον προσδιορισμό έδρας. Όχι για την ίδια την έδρα, αλλά τον προσδιορισμό μιας έδρας, πώς θα γίνεται. Θεωρώ κατά τα άλλα ότι εδώ σε αυτό το σημείο δεν θα πρέπει να μιλήσουμε για μετεγκατάσταση αυτής της ε, υπηρεσίας. Είμαι υπέρ του να παραμείνει η έδρα στην Ελλάδα, όπως το αποφάσισε το Συμβούλιο εξάλλου και σε σύμφωνη γνώμη με την Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση. Η κυρία Ποδηματά από πλευρά τη θα μπορέσει να διοργανώσει μια συνάντηση μεταξύ εισηγητών, σχεδόν εισηγητών και εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης για να εξεταστούν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή ποια κριτήρια υπάρχουν και ποιες δυνατότητες υπάρχουν τελικά που προσφέρονται από την ευρωπαϊκή κυβέρνηση στο θέμα της έδρας να, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και να επιληθεί. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχει ήδη μια ομάδα εργασίας που ασχολείται με αυτά τα θέματα της αξιολόγησης δηλαδή της αποτελεσματικότητας όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών και υπηρεσιών. Τώρα ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας αν πούμε γιατί αυτή η υπηρεσία να έχει αυτή την έδρα και όχι άλλη. Και είναι σκόπιμο να γίνεται αυτό ή όχι. Πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να παραμείνει σε αυτή την έδρα η ΕΝΗΣΑ και να εξετάσουμε περισσότερο το θέμα πώς μπορεί να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ε, υπηρεσίας. Δεν χρειάζεται διευρυμένη εντολή. Ο κύριος Τσουκαλάς παρακαλώ. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, όπως σας είχα υποσχεθεί, σας έχω στείλει μια λεπτομερή επιστολή για να αντιμετωπίσω τα τεχνικά ζητήματα. Θα εστιαστώ ο κύριος Σέλερ και η κυρία Τικάου με μεγάλη ε, ευκρίνεια έθεσαν τα κύρια ζητήματα του ΕΝΙΖΑ. Το πρώτο ζήτημα του ΕΝΙΖΑ είναι τι σόι ΕΝΙΖΑ θέλουμε. Ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός. Κάτι δική μου αντίληψη ο ΕΝΙΖΑ πρέπει να έχει αυξημένο διεθνή ρόλο και αυξημένη ορατότητα τόσο σε σχέση με τους διεθνείς οργανισμούς που εμπλέκονται σε θέματα διαδικτύου όσο και με τους διεθνείς μας εταίρους. Πρέπει να αποτελεί το single point of contact για ό,τι έχει να κάνει με κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη. Από τα ζητήματα που ετέθησαν ήταν το ζήτημα του mandate. Θεωρώ ότι η πρόταση της κυρίας Τικάου είναι πολύ λογική. Θα έπρεπε να υπάρχει permanent mandate με αξιολόγηση κάθε πέντε χρόνια έτσι που να μπορούμε να κάνουμε τις αναγκαίες τροποποιήσεις όπως ο κύριος Έλερ ε, προδιέγραψε. Ένας λαθρεπιβάτης της συζήτηση υπήρξε το ζήτημα του location. Ούτε κατά αρμοδιότητα, ούτε κατά εντολή υπήρξε ζήτημα της έδρας στο ε, report αυτό δεν αντιλαμβάνουμε πλήρως την ε, επιμονή που έχει να κάνει με τη location και την αποτελεσματικότητα του ΕΝΙΖΑ. Αντιθέτως, ο κύριος Σωσή, που ήταν αυτός που έκανε την αξιολόγηση από το Court of Auditors, ήταν ιδιαίτερα σαφής σχετικά με το πρόβλημα του ΕΝΙΖΑ. Μας είπε ότι ο ΕΝΙΖΑ είναι ένα από τα μικρότερα ευρωπαϊκά agencies με λιγότερο από 60 άτομα προσωπικό. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τις όποιες διοικητικές δυσλειτουργίες παρουσιάζει. Το πρόβλημα του Ενίζα δεν είναι ότι βρίσκεται μακριά. Το πρόβλημα του Ενίζα είναι ότι είναι μικρός και οφείλουμε να τον ενισχύσουμε. Θεωρώ επίσης ότι με τον Ενίζα και την αμφιθυμία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το ρόλο του επαναλαμβάνεται ο χορός σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Αυτή τη φορά δεν έχουμε να αποφασίσουμε για το ποιο θα είναι το ευρώ και η κοινή οικονομική πολιτική, αλλά ποιος θα είναι ο ρόλος του ΕΝΙΖΑ σε μια Ευρώπη άλλης μορφής που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να είμαστε αποφασισμένοι να συζητήσουμε. Και με την ευκαιρία αυτή και τελειώνω, καλά θα ήταν το Ευρωκοινοβούλιο αντί να ασχολείται με own initial reports να ασχοληθεί επιτέλους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 ε, υπάρχουν πιέσεις για να πάρουμε μέτρα πιο αποτελεσματικά στον τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου. Έχουν ξεκινήσει ορισμένα προγράμματα και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς δεν μπορούμε να επωφεληθούμε την εμπειρία που έχει το ΝΑΤΟ στο συγκεκριμένο τομέα και θέλουμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν, να κάνουμε αναγκαστικά λάθη και να αναγκαστούμε τα λάθη αυτά να τα αποκαταστήσουμε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται το θέμα. Η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 10 Νοεμβρίου. Ακολουθούν τώρα οι ψηφοφορίες. Όλοι ελπίζω έχετε τις κάρτες σας. Ξέχασα να ρωτήσω αν, έχετε, αν εγκρίνετε τα πρακτικά της 8ης Σεπτεμβρίου. Ωραία λοιπόν. Τότε... περνάμε έτσι στις ψηφοφορίες αφού εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη έχουμε που πρέπει να ψηφίσουμε σχετικά. Λειτουργούν οι συσκευέ σα, ναι. Είναι Λειτουργούν οι συσκευέ. Πρώτο σημείο. την, την πολιτική γειτονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε τα χαρτιά στη διάθεσή σας. Περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβιβασμός 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 5. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε το 9 υπέρ κατά αποχές κάποιες ψήφοι εναντίον εγκρίθηκε 10 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 17 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε στην τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα εγκρίθηκε να δω πάλι υπέρ 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 31 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 31 τροπολογία. 31. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα 37 συμμετείχαν, 19 εναντίον. Εσείς είσαστε υπέρ ή εναντίον. Υπέρ. 18-19 το αποτέλεσμα. 19 εναντίον, 18 υπέρ. Απορρίφθηκε. 36 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 47 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 6 συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 60 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και τώρα θα ψηφίσουμε τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία τελική ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας τώρα και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Θερμά συγχαρητήρια κύριε συνάδελφε. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Ψήφισμα. Η ουδετερότητα στα δίκτυα. Και εδώ έχουμε ένα πίνακα έχετε χαρτιά στα χέρια σας. Ελπίζω να έχουμε προχωρήσει. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 1. Όχι. Τροπολογία 2. Και ΙΜΚΟ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν συμβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμό όχι τροπολογία 6 συγγνώμη με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 45 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 46 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά Αποχέ εγκρίθηκε. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 61 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ΙΜΚΟ παράγραφος 4 στην παράγραφο 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Στο τέλος ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Τι ξέχασα είπατε, τι λέτε. Χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεται. 46 ξέχασα, όχι, την, την ψήφισα. Περνάμε στην συνολική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Και τώρα, ναι, αργά αργά Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και εγκρίθηκε. Ομόφωνα κιόλας εγκρίθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά εισηγητά. Και έτσι... Ναι, όλα έχουν τις επιπτώσεις τους. Πρέπει να ευχαριστήσουμε κάθε εισηγητή ένα προς ένα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές, διότι ήταν πολύ δύσκολο με το ψήφισμα να ευρεθεί μια συμφωνία. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Αλλαγή της οδηγίας για την αναθεώρηση των κοινών διατάξεων πλαισίου για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων και τη φορολογία τους. Ο συνάδελφος Κόβατς ως πρώτος και μόνος θα παρέμβει. Πού είναι ο κύριος Κόβατς? Συνάδελφε Κόβατς έχετε τον λόγο. Τους άλλους συναδέλφους παρακαλώ για άλλη μια φορά. Αν έχετε κάτι πολύ σημαντικό το οποίο κατανοώ να συζητήσετε, να βγείτε εκτός αιθούσης. Εντάξει. Αυτό είναι όχι μόνο σε σχέση με τα μέλη, αλλά και για τους βοηθούς, τους φιλοξενούμενους. Αν θέλετε να συζητήσετε, εκτός αιθούσης παρακαλώ. Είναι δίκαιο και ε, φιλικό και ευγενές προς τους, προς ε, συμμετέχοντες. Ο κύριος Κόβατς, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι όσον αφορά την ενεργειακή αυτή οδηγία για το, το 2003 96 ε, ΟΚ οδηγία δηλαδή που πρέπει τώρα να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ο γενικός στόχος ποιος είναι είναι η φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων να αναδομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήξουμε σε, μια, σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα βιομηχανία και παραγωγή ενέργειας και να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όσον αφορά το περιβάλλον. Οι διαφορετικές ενεργειακές πηγές να τύχουν ίσης αντιμετώπισης, δίκαιας αντιμετώπισης και να δημιουργηθεί ένα γενικό πλαίσιο για την φορολόγηση των διαφορετικών ενεργειακών προϊόντων ή τη φορολόγηση, α το πω έτσι, του διοξιδίου του άνθρακα που εκλείεται κατά την παραγωγή. Γι' αυτό η ελάχιστη φορολόγηση θα πρέπει να ε, μπορέσει να διαρρεθεί με τέτοιο τρόπο ένας φόρος που θα είναι ο φόρος που θα αφορά το διοξίδιο του άνθρακα 20 ευρώ ανατόνο ε, διοξιδίου του άνθρακα η άλλη μορφή φορολογίας θα είναι ε, η γενική φορολόγηση ενέργειας ή ενεργειακών προϊόντων που θα αφορά το περιεχόμενο ενέργειας ε, που ε, οδηγούμε στο να επιτυγχάνουμε από την χρήση των πρώτων υλών. Χαιρετίζω τις προτάσεις ε, για την ε, αναθεώρηση αυτής της οδηγίας πλαισίου για τη φορολόγηση. Ιδιαίτερα, μια και η οδηγία αυτή θα μπορεί να συνάδει με τους στόχους ε, της προστασίας του περιβάλλοντος και τις πολυσχηδείς, τους πολυσχηδείς στόχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά θέλω να τονίσω πόσο σημαντική θα είναι η οδηγία αυτή μια και το ότι μέχρι σήμερα τα ίδια τα κράτη-μέλη καθόριζαν ποιο θα είναι το ενεργειακό μείγμα. Εξάλλου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις αυτή η οδηγία στην οικονομία γενικά όσον αφορά τις εταιρείε και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενεργειακά και γι' αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί να διευκρινιστεί άμεσα πώς θα διαμορφωθεί η νομική βάση ως προς αυτά. Και σε σχέση με τις ε, μελέτες επιπτώσεων και με λεπτομερείς ή εξειδικευμένες παρατηρήσεις που θα διασφάλιζαν ότι θα βρίσκεται σε ευθυγράμμιση, θα συμμορφώνεται αυτή η οδηγία με την αρχή της επικουρικότητας για τον τομέα της ε, κοινής συναρμοδιότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την πτυχή αλλά επίσης και τις διαφορετικές, τα διαφορά μέτρα τα οποία θα καθοριστούν που θα πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά για στους πολίτες και να είναι πιο αποτελεσματικά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει εξειδικευμένα σε λεπτομέρειες και με σαφήνεια να τεκμηριώνεται πάντα γιατί χρειάζεται αυτή η οδηγία ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να κατανοήσουν, να είναι εύληπτο για τους πολίτες πώς θα δράει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα και γιατί θα πρέπει να δράμε με αυτόν τον τρόπο. Οι διάφορες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις ε, είναι επίσης σημαντικές και πρέπει να μας κάνουν να ανησυχούμε. Κατά πρώτο λόγο, μέσω των διαφορετικών αυτών μέτρων που προβλέπονται από την οδηγία, δεν υπάρχει σε βάθος επαρκής ανάλυση ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, που θα συνεπάγεται αυτή η οδηγία για τα επιμέρους κράτη-μέλη. Πέρα από αυτό όμως θα έπρεπε ευέλικτες λύσεις να επιτευχθούν, να προταθούν ευέλικτες λύσεις ως δυνατότητες και θα μπορούσαν και μεταβατικές περίοδοι να καθοριστούν πράγμα που ίσως θα ήταν αναγκαίο. Η βιομηχανική πολιτική παραμένει εκτός όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η βιομηχανική πολιτική. Μια κοινή φορολογική βάση όσον αφορά την σύσταση των ενεργειακών προϊόντων ήδη στα κράτη-μέλη θα συνεπάγεται αλλαγή της φορολογικής βάσης και από πλευρά των κρατών μελών είναι σημαντικό να υπάρχει μια μελέτη επιπτώσεων για όλου του βιομηχανικού τομεί ω προ αυτά, ώστε η ανταγωνιστικότητα από πλευρά Ευρώπη να μπορεί να διασφαλιστεί. Κατά την επανεξέταση τη ε, οδηγία αυτή για τη φορολόγηση, δεν επιτρέπεται να καταλήξουμε ότι, ώστε να υπάρξουν στρεβλώσεις στην αγορά και να χάσουμε ενδεχομένως θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον θα πρέπει και με τους άλλους τομείς πολιτικών να ε, συνάδουν οι προτάσεις αυτές. Την τελευταία φορά το 2003 καθορίστηκαν τα ποσοστά και τα όρια φορολόγησης ε, σε αυτόν τον τομέα. Και εγώ πιστεύω ότι μια επανεξέταση χρειάζεται ώστε να ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός και άλλοι παράγοντες και επιπλέον να εξεταστούν και οι οικολογικές επιπτώσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη των διαφορετικών καυσίμων και γι' αυτό χρειάζεται ένα ενιαίο πλαίσιο όμως μέσω μιας αυτόματης ε, τιμαριθμικής προσαρμογής θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη το ύψος αυτών των, ε, τον καθορισμό αυτό να τον ε, απολέσουν τα κράτη-μέλη ως αρμοδιότητα και φοβούμε ότι σε σχέση με τον καθορισμό αυτών των ορίων ίσως θα μπορούσαν να ανέβουν πολύ, να αυξηθούν πολύ αυτές οι τιμές και αυτό θα μπορούσε να έχει άμεσα αρνητικές επιπτώσεις, κοινωνικά αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τις υψηλές τιμές στις οποίες θα καταλήξουν. Λίγαμε για τους τελικούς καταναλωτές, τους ε, καταναλωτές γενικά. Μια, ένας, μια αυτόματη αναπροσαρμογή θα μπορούσε να αποτελεί μια δυσανάλογη επιβάρηση ε, εις βάρος των καταναλωτών. Επίσης θα ήθελα να πω ότι οι τιμές καυσίμων τα προηγούμενα ε, χρόνια αυξήθηκαν ήδη σημαντικά και κατά τα άλλα επιπλέον οι τιμές θα μπορούσαν και για τα ενεργειακά προϊόντα και για τα καύσιμα όσον αφορά την γεωργία και την δασοκομεία να δούμε ότι ίσως θα μπορούσαν να αυξηθούν πάλι οι τιμές. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση τις εθνικές δομές φορολόγησης να τις καθορίζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στον τομέα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και την έκκληση διοξιδίου του άνθρακα πολλές επενδύσεις, μεγάλες επενδύσεις ε, απαιτούνται να γίνουν και γι' αυτό είναι σημαντικό στην φορολόγηση του ντίζελ και της βενζίνης ε, ως καυσίμων να πετύχουμε ότι θα υπάρχουν κίνητρα για την χρήση του ντίζελ και η φορολόγηση του ντίζελ δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη από εκείνη της ε, βενζίνης. Θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω οπωσδήποτε πρώτα τη γραμματεία της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής κατά τα άλλα επίσης και τους συναδέλφους που με βοήθησαν να συντάξω αυτή τη γνωμοδότηση από πλευράς μου. Και θα ήθελα να προσθέσω κιόλα εδώ ότι θα ήθελα να πω ότι η κυρία Άστριτ Λούλινγκ παρόμοια θέση υιοθετεί όπως και εγώ όσον αφορά τις απόψεις της και ευχαρίστω έτσι με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και αυτή. Η κυρία, ο κύριος Γκλάντε παρακαλώ. <coughs> Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου κάποιε παρατηρήσει να κάνω για αυτή την οδηγία για την ενεργειακή ε, φορολόγηση εκ μέρου συναδέφου που δεν μπορεί τώρα σήμερα να παραστεί εδώ. Η ομάδα μας χαιρετίζει την αναθεώρηση της ενεργειακής αυτής οδηγίας και ζητούσε και εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα μια φιλόδοξη αναθεώρηση της φορολόγησης αυτής στην οδηγία που έχει επιτευχθεί ήδη από το 2003 θα πρέπει να προσαρμοστεί προς τους περιβαλλοντικούς στόχους και πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν και κίνητρα για τη μείωση έκκλησης διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει επιπλέον να επιτυγχάνεται η προώθηση των επενδύσεων, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας αντανακλά σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ανάγκες και συνιστά ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Οι παράγοντες κλειδιά είναι σαφείς και λογικοί. Το θέμα των καυσίμων είναι επίμαχο. Αλλά η κυρία Βόρσκοπ νομίζει ότι όλα τα καύσιμα για τους κινητήρες και για τη θέρμανση με ουδέτερο τρόπο αμερόλητα πρέπει να φορολογούνται και κριτήριο θα πρέπει να είναι το ποσοστό διοξιδίου του άνθρακα που εκλείεται. Να επιβραδύνω πρόεδρε. Ένα, ένα πρόβλημα ίσως θα υπήρχε και εδώ ναι, ελπίζω ότι κατάφεραν οι διερμηνείς να παρακολουθήσουν ε, εκ μέρους της ε, κυρίας συναδέφου εκφράζω αυτές τις απόψεις. Έχει νόημα να υπάρχει ένα ισοδίκαιο πλαίσιο λοιπόν όσον αφορά τον ETS, τομέα ETS και εκτός ETS. Ένας φιλόδοξος στόχος για την οδηγία αυτή θα πρέπει να είναι να συνεισφέρουμε στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και στην δημιουργία θέσεων πράσινης απασχόλησης όπως αποκαλείται όσον αφορά φιλοπεριβαλλοντικές δηλαδή θέσεις απασχόλησης. Να μην ξεχνάμε και τα κράτη-μέλη της <clears throat> ε, εκπομπές ρήπων θα πρέπει μέσα σε ένα ξεχωριστό νομικό πλαίσιο να τις ρυθμίζουν ως αποτελεσματικό μέσο ε, για τη διαμόρφωση του κόστους θα πρέπει να λειτουργήσει και η οδηγία αυτή θα πρέπει να είναι ένα σωστό μέσο να ενδυναμώσουμε την αποτελεσματικότητά μας σε αυτή την πολιτική. Δεν έχει δυστυχώς το Ευρωκοινοβούλιο δυνατότητα συναπόφασης εδώ. Πρέπει όμως υπεύθυνα να δράσουμε και να δείξουμε ότι την πρόταση της Επιτροπής στον πυρήνα την υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Βασιλεύει η Βασιλεύει σύγχυση. Θα συνεχίσω λοιπόν μετά από αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι Ούσκορ και Γκλάντε. Υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία καθιστά πιο συνεκτική την διαδικασία φορολόγησης της ενέργειας αλλά διασφαλίζει και τη συμβατότητα ανάμεσα στη συγκεκριμένη πολιτική και στην πολιτική προστασία του κλίματος. Θέλουμε λοιπόν το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει γενικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν κατάλαβα καλά, η Επιτροπή μας έχει παράδοση, θα έλεγα, να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της βιομηχανίας και το κατανοώ αυτό, αλλά για ποια βιομηχανία μιλάμε. Μιλάμε για τις παλαιού τύπου βιομηχανίες ή θέλουμε να προωθήσουμε τις ε, μελλοντικές, τις βιομηχανίες του μέλλοντος μάλλον. Φοβάμαι ότι συνήθως κοιτάμε πίσω και όχι μπροστά. Και μάλιστα βρήκα τον τόνο του εισηγητή πάρα πολύ αμυντικό, αδικαιολόγητα αμυντικό λέει ότι δεν ξέρουμε που πάμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Πρέπει να πρασπιστούμε τα συμφέροντα των κατών μελών. Πρέπει να προστατεύσουμε από κοινωνικέ επιπτώσει. Για κοιτάξτε λίγο, στον τομέα της φορολογία της ενέργειας γνωρίζουμε ήδη ότι η ενέργεια δεν είναι κάτι μόνο που συνιστά μια παγκόσμια αγορά, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη όταν μιλάμε για τη μεταφορά προφανώς της ενέργειας μιλάμε για διασυνοριακές δραστηριότητες και κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε αυστηρά εθνικό επίπεδο. Και όταν λέμε, όπως λέει ο εισηγητής, δεν πρέπει να στερήσουμε από τα κράτη-μέλη την δυνατότητα να φορολογήσουν σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερο να έχουμε κοινωνική φορολογία, κοινοτική φορολογία και όχι εθνική φορολογία και δεν πρέπει να είμαστε εθνικιστές στον συγκεκριμένο τομέα. Για την κοινωνική πλευρά, την υπογραμμίζω πράγματι αυτή την πλευρά όταν αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας και πράγματι αυξάνονται, υπάρχουν κοινωνικές επιπτώσεις τις οποίες καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη όμως δεν θα πρέπει εμείς με ένα μέτρο να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις συνέπειες της αύξησης της τιμής στις πιο ευάλωτες ε, πλευρές, στα πιο ευάλωτα κομμάτια του πληθυσμού κάποια κράτη-μέλη, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και άλλα κράτη-μέλη, τα οποία πράγματι εφαρμόζουν τέτοιου είδους γραμμικούς φόρους, αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στους οικονομικά ασθενέστερους. Αυτές οι χώρες λοιπόν μας λέτε κάντε προσέξτε γιατί θα πρέπει να θίξετε τους πιο ευάλωτους. Εγώ θα ήθελα να καλέσω τα κράτη-μέλη πρώτα να εφαρμόσουν ή να εφαρμόσουν σωστά ή να εφαρμόσουν με ποσοστά την φορολογία τους και όχι να λέτε ότι έχουμε πρόβλημα υπερασπιζόμενοι τους κοινωνικά ασθενέστερους, τους οικονομικά συγγνώμη ασθενέστερους. Είμαι εισηγητή και στην ΕΚΟΝ. Δεν πρέπει να λέμε τα ίδια πράγματα σε όλε τι επιτροπέ, αλλά νομίζω ότι κάθε επιτροπή πρέπει να συγκεντρώνει την προσοχή τη στον τομέα τη. Πρώτον, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την κυροζήνη, το καύσιμο των αεροσκαφών και τα καύσιμα για την κίνηση των πλοίων. Και αυτό λέει και η πρόταση τη Επιτροπή και πρέπει να το δεχτούμε η εξαίρεση της κυροζήνης από τη φορολογία είχε συμβεί την εποχή που θέλαμε να καταστήσουμε τις αερομεταφορές πιο προσβάσιμες σε όλους. Τώρα όχι μόνο είναι προσβάσιμες οι αερομεταφορές, αλλά είναι υπερβολικά προσβάσιμες και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα και να φορολογήσουμε επιπλέον τα καύσιμα των αεροσκαφών. Τώρα για την τεχνική ουδετερότητα της φορολογίας. Μπορώ να μπω σε μια τεχνική συζήτηση για τον ντίζελ, αλλά θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνον το ότι το ντίζελ μπορεί, μπορεί να είναι ή μπορεί και να μην είναι εντατικό σε επίπεδο διοξίδιο του άνθρακα αλλά παράγει μόλυνση, προκαλεί μόλυνση και σε άλλους ε, τομείς. Ξέρουμε τι γίνεται με τα λεπτά σωματίδια και την παραγωγή τους από την καύση δίζελ. Λοιπόν, ε, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Επίσης να γνωρίζουμε πρέπει ότι υπάρχει μια τάση επιστροφή στη βενζίνη και όχι αιμονή στο πετρέλαιο για την κίνηση, την αυτοκίνηση. Και σύν της άλλης θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα καταστούμε λιγότερο εξαρτημένοι σε καύσιμα από ό,τι σήμερα. Και τέλος για τον εισηγητή. Υπάρχει κάτι το οποίο με ανησυχεί. Γνωρίζουμε ότι η τελευταία συζήτηση και απόφαση για τη φορολογία στην ενέργεια χρειάστηκε πέντε χρόνια για να προχωρήσει. Όταν το κοινοβούλιο αυτό δίνει την εικόνα της κολυσιεργίας όταν επιβραδύνει τις εξελίξεις στην Ευρώπη, σίγουρα υπό τις παρούσες συνθήκες προσφέρουμε κάκιστη υπηρεσία στην Ευρώπη. Είναι μια τακτική την οποία μερικές φορές μπορώ να κατανοήσω, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Το κοινοβούλιο αυτό έχει δείξει ότι θέλει να δουλέψει γρήγορα αποτελεσματικά και να κλείσει θέμα αν είναι θέματα αν είναι δυνατόν και στην πρώτη ανάγνωση. Επιτρέψτε μου ε, να κάνω την εξής παρατήρηση. Κάθε επανεξέταση δεν σημαίνει απαραίτητα καθυστέρηση. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός. Οι διαδικασίες είναι ήδη αρκετά δυσχερείς και ο χρόνος ε, που είναι απαραίτητος πρέπει να διατίθεται. Κύριε κυρία Τσικάου. Πέντε ώρα θα σταματήσω. Κύριε Τικάου. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ στη μέσα ανατόνο διοξιδίου του άνθρακα, έκκλησης διοξιδίου του άνθρακα. 20 ευρώ ανατόνο εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα αναφέρονται στο παράτημα. Γνωρίζω ότι το ETS, το πακέτο μέτρων εκπομπής ρήπων, και με άλλες τιμές 33 ή 13 ευρώ είχε προταθεί. Γι' αυτό θέτω κάποιες ερωτήσεις. Είναι ίσως κάπως αυθαίρετο 20 ευρώ τόνο να καθορίζεται για τις ενεργές μεταφορές και σύμφωνα με την οδηγία FCC προστασίας του κλίματος θα έπρεπε οι εναερίες μεταφορές από το 2012 συμπεριλαμβάνονται στις εκπομπές ρήπων. Επιπρόσθετη δηλαδή φορολόγηση της κυροζήνης θα σημαίνει αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά πρακτικά διπλή φορολόγηση όσον αφορά τις εναερίες μεταφορές. Αν τώρα γίνεται συζήτηση και όταν γίνεται συζήτηση για τους θεσμούς και τις προβλέψεις και τα όσα θα υπάρχουν στο πακέτο αυτό, και δεν θα είναι μόνο μια φορολόγηση προσωρινή ή μεταβατική, ε, τότε πιστεύω ότι και οι εναέριες μεταφορές θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το πλαίσιο. Και μια τελευταία παρατήρηση τώρα οι ενεργειακές τιμές που αφορούν τους τελικούς καταναλωτές και που εκείνοι θα πληρώνουν. Τα ιδιωτικά νοικοκυριά κυρίως έχω υπόψη μου. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να διαρωτηθούμε ποια μέτρα είναι εκείνα τα οποία μπορούμε να αναλάβουμε ώστε όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά πραγματικά υπό αξιοπρεπείς συνθήκες να μπορούν να, ζουν ώστε να μην υπάρχει ενεργειακή παινία ή φτώχεια. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Δεν νομίζω να υπάρχει κίνδυνος να με συγχύσετε με κυρία. Από τη σκοπιά λοιπόν του Λαϊκού Κόμματος, σε ό,τι αφορά τη νέα διάρθρωση των ελαχιστών φορολογικών συντελεστών, εγώ η αύξηση αυτή φαίνεται να οδηγήσει σε μείωση ε, της αγοράς δίζελ κατά 30% και είναι και σε αντίθεση με την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης. Δεν μπορούμε ως Ευρώπη από τη μια μεριά να βάζουμε αυστηρά όρια για τα εκπαιμπόμενα οξύδια του άνθρακα και να ζητούμε μηχανές οικονομικές σε κατανάλωση και μετά να ερχόμαστε να υπερεπιβαρύνουμε με φορολόγηση αυτό το καύσιμο το οποίο είναι πιο οικονομικό σε κατανάλωση δηλαδή. Όλες οι επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα ε, στην, ε, ε, στον εξυγχρονισμό, μάλλον στη, στην έρευνα για, τέτοιες, για τέτοιους κινητήρες πηγαίνουν περίπατο. Ανατρέπεται δε και η ισορροπία ανάμεσα στις φορολογήσεις των διαφόρων ε, παραγόντων. Γι' αυτό είμαστε αντίθετοι με αυτήν την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε αυτό να είναι και το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τους Υπουργούς. Η κυρία Γιόρδαν Σίσελη. Ρωμάνα Ζόρδαν Σίσελη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντοτε τάχθηκα υπέρ ενός σαφούς καθορισμού των στόχων μας και βέβαια τις προσπάθειες επιδιώξης σε όλα τα επίπεδα. Και στο παρόν έγγραφο βλέπω κάποια θετικά στοιχεία. Αφού πρόκειται για σημαντικό στόχο, δηλαδή να ληφθούν υπόψη και τα περιβαλλοντικά προβλήματα σε σχέση με την φορολογική πολιτική. Μέχρι τώρα δεν είχαμε πολλή σχέση με φορολογική πολιτική, ιδίω στην παρούσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Γι' αυτό θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της αναθεώρησης. Δεν θα ήθελα βέβαια να καθυστερήσει η προσπάθεια αυτή αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε επαρκεί πληροφορίε για να μπορούμε να κρίνουμε πού βρισκόμαστε και προ τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε και ποιε όπω είπα θα είναι οι επιπτώσει τη νομοθετική αυτή πρόταση. Εγώ βλέπω εδώ ελλειπή πληροφόρηση, δηλαδή δεν βλέπω κάποια στοιχεία που να λένε πώς θα λειτουργήσει το σύνολο του συστήματος. Εξήγησαν με ποιον τρόπο διασυνδέεται το σύστημα με τις εναέριες μεταφορές, αλλά πώς θα λειτουργήσει, ποιες θα είναι οι διάφορες εντός εισαγωγικών συνέργειες, δεν το γνωρίζουμε. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι τα αποτελέσματα του, της χρήσης του ενός συστήματος, του άλλου, γιατί χρειαζόμαστε το ένα ή το άλλο, πώς συνδέεται η χρήση των συστημάτων. Περισσότερες πληροφορίες λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή. Και όπως διαπιστώνει ο εισηγητής, αυτό θα οδηγεί σε περαιτέρω επιβαρύνσεις και των τιμών του φυσικού αερίου. Είπαμε πρόσφατα ότι 3 δισεκατομμύρια από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πρόκειται να διατεθούν για το αέριο. Δηλαδή με το ένα χέρι δίνουμε, με το άλλο χέρι παίρνουμε. Και εν πάση περιπτώσει επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε επαρκή ενημέρωση για τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Κύριε Κόβατς, επιθυμείτε να επανέλθετε. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Θα τροποποιήσω το κείμενό μου σύμφωνα με τις προτάσεις που εκφράστηκαν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο στην ημερησία διάταξη. Να επισημάνω ότι στις 9 Νοεμβρίου το μεσημέρι θα έχουμε την κατάληξη της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών. Εντάξει, περνάμε στο επόμενο σημείο. Ενεργειακή ε, αποδοτικότητα και σε σχέση με τις οδηγίες. Έχουμε ξανασυζητήσει, θα ήθελε τώρα μέχρι τις και μισή έχουμε χρόνο. Θα ήμουν ευγνώμος ευγνώμων επειδή πάρα πολλοί θέλουν να παρέμβουν. Παρακαλώ να είσαστε σύντομοι γιατί δεν θα τα καταφέρουμε αν μακρηγορήσετε. Είναι σημαντική προϋπόθεση για την εξέλιξη των εργασιών μας. Ήδη προανέφερα η κατάληξη της προθεσμίας θα είναι στις 7 το βράδυ, τα μεσάνυχτα 24.00. Θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε σε σχέση με τα θέματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρέπει τις προτάσεις να εξεταστούν. Ο κύριος Τούρμες έχει πρώτος τον λόγο. Παρακαλώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Λοιπόν, και πάλι κάποιες έννοιες, κάποια σημεία σύντομα. Και στο τέλος, αν θα υπάρχει χρόνος, θα μπορούσα να ανταποκριθώ στις παρεμβάσεις των συναδέλφων που θα έχουν γίνει. Εδώ έχουμε το θέμα της κλιματικής πολιτικής αλλά και της οικονομικής πολιτικής. Δίνουμε δισεκατομμύρια για να αγοράσουμε πετρέλαιο εκτός Ευρώπης. Αν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην Ευρώπη, αν θέλουμε να έχουμε περισσότερα κονδύλια στην Ευρώπη για πρόσθετη αξία και θέσεις απασχόληση, πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αν θέλουμε να αποφύγουμε <clears throat> τις επόμενες δεκαετίες όπου θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τα, συστήματα, τα ενεργειακά συστήματα και να έχουμε επενδύσεις καλό θα ήταν αυτή η οδηγία που θέλει να προωθήσει την αποδοτικότητα της ηλεκτρικής ενέργειας γιατί θα χρειαζόμαστε λιγότερα καλώδια, λιγότερες, ε, λιγότερους ε, σταθμούς παραγωγής. Το ουσιαστικό μας πρόβλημα είναι πώς αυτά τα κονδύλια, αυτές οι δράσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αυτές οι επενδύσεις θα επιτευχθούν, πώς θα εξευρεθούν αυτά τα κονδύλια, πώς βράχει πρόθεσμα θα καλυφθούν οι ανάγκες. Γι' αυτό ένα ξεχωριστό άρθρο, μια ξεχωριστή παράγραφο συντάσσω που προβλέπει την γεφυροποίηση, την δυνατότητα συνδυασμού με τις προτάσεις ε, του Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική Συνοχής, αλλά και project bonds ομόλογα έργων. Γιατί να μην μπορούν και αυτά να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Ή τα κονδύλια, για παράδειγμα, από τις εισπράξεις όσον αφορά την έκκληση διοξιδίου του άνθρακα έσοδα από το 2013 και εφ' Και για την κτηριακή πολιτική όχι μόνο για τα δημόσια κτίρια πρέπει να συζητήσουμε αλλά συνολικά να οδηγηθούμε σε ένα οδικό χάρτη, ένα δρομολόγιο για τα κτίρια. Είμαι υπέρ του, της εξισορρόπησης ε, των αγορών και όσον αφορά και τη ζήτηση διότι και στι είπα θα είναι πιο φθηνή η παραγωγή, όχι μόνο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η αποδοτικότητα και θα μειωθούν οι τιμές και θα μπορούν να μειωθούν οι τιμές ώστε να εξισορροπηθούν οι αγορές ε, όσον αφορά αυτή την πτυχή. Είμαι υπέρ της ε, μεγαλύτερης εμπλοκής των καταναλωτών και έχω και σε σχέση με κάποια σημεία που έχει το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάποιες βελτιώσεις. Ε, ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τώρα να συνεχίσουμε με τον κατάλογο. Α ξεκινήσουμε με τον κατάλογο. Σκιώδης εισηγητές πρώτα. Οι εκπρόσωποι του Πίπερ, συνάδελφος Πίπερ πρώτος, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η οδηγία είναι πράγματι σημαντικό βήμα. Προσφέρει κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και επομένως μείωση της εξάρτησής μας. Ταυτόχρονα είναι και σημαντική η συμβολή της για την προστασία του περιβάλλοντος και για μια όθηση προς ε, νέα μέσα παραγωγής ενέργειας που να είναι λιγότερο ε, που να είναι πιο οικονομικά. Ο κ. Τούρμας έχει κάνει σχετικές τροπολογίες και υπάρχουν ορισμένε ιδέες με τις οποίες θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε για τις οποίες θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν μπορούμε να βάλουμε βέβαια στο ίδιο καλάθι όλες τις ε, χώρες, ενώ το burden sharing, καθώς και οι άλλες ιδέες του είναι ενδιαφέρουσες. Τώρα, βέβαια, η οδηγία θα ήταν καλύτερη εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε περιοριστεί να θέσει μόνο ορισμένες συνθήκες πλαίσια, διότι τώρα μπαίνει σε υπερβολικές λεπτομέρειες, κάτι που ε, για μας μπορεί να ρυθμιστεί καλύτερα στο εθνικό επίπεδο η οδηγία θα ήταν ακόμη καλύτερα βέβαια, ακόμη καλύτερη, εάν περιλάμβανε έναν ενιαίο ορισμό της αποδοτικότητας της ενέργειας, που δεν το κάνει, αλλά το κάνει ο κ. Τούρμες. Ε, αποδοτικότητα της ενέργειας ίσον εξοικονόμηση ενέργειας, λέει. Τελεία. Κατά τα άλλα, η έκθεση του συναδέλφου ε, λέει όχι διπλού επίπεδου προσέγγιση, ε, να μην υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση, περαιτέρω υποχρεώσεις κοινοποιήσεως κλπ. Εγώ νομίζω ότι μάλλον βρίσκομαι λίγο αμήχανος μπροστά σε όλες αυτές τις ε, προτάσεις για να γίνει πιο αυστηρό το κείμενο. Για παράδειγμα, για την συμπαραγωγή ενέργειας, εάν δεν είναι οικονομικά τα κριτήρια της εφαρμογής τους στις ε, περιφέρειες, τότε μπορούν να υπάρξουν και εξαιρέσεις στις χώρες μέλη. Ολόκληρη αυτή την παράγραφο προτείνει η συγκητής να τη διαγράψουμε με την απλή αιτιολόγηση ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να υποφελούνται από τη συμπαραγωγή και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει λόγος να γίνουν εξαιρέσεις. Εμένα μου φαίνεται υπερβολικά ε, σκληρό το επιχείρημα αυτό, αγαπητέ συνάδελφε, και διαρωτώ με αν θα μπορέσουμε έτσι να συμφωνήσουμε. Για τα άθα τώρα επιμέρους, επειδή ο κύριος Τούρμες έχει περιγράψει έτσι αυτό το νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό, εγώ θεωρώ ότι βασίζεται, βασίζεται σε κλειδονιζόμενη βάση. Και για το άρθρο 6 που λέει ότι θα τροφοδοτείται από ε, πρόστιμα και για τα μικρότερα μέτρα τα οποία επιθυμούμε να προτείνουμε εμείς περισσότερο για μικρές ε, κοινότητες Υποτίθεται ότι τροφοδοτείται και από τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα διαρθρωτικά ταμεία όμως είναι ευθύνη των χωρών μελών και 50% συγχρηματοδότηση, για παράδειγμα στην περιφέρειά μου, 50% θα πρέπει δηλαδή να αναλάβουν το 50% οι ε, τοπικές κοινότητες και σε ένα μέρος από, από ε, κονδύλια της Ευρωπαϊκής ε, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι όμως περίπλοκα αυτά. Εμείς νομίζουμε ότι χρειάζεται καλύτερα να μεταφέρουμε τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που έχουν αποδείξει την αξία τους. Μην προχωρείτε όμως, μην προχωρήσει όμως το κείμενο σε λεπτομερή ε, απαρίθμηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τις χώρες μέλη. Για το άρθρο 3 νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει η διεπίπεδη αυτή προσέγγιση, διότι χρειαζόμαστε πολλά ε, πολλά πράγματα ακόμα και η οδηγία eco-design πρέπει και αυτή να αποδείξει εάν λειτουργεί και πιστεύουμε επίσης ότι η υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας με κανένα τρόπο δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Αν λοιπόν κάποιες χώρες μέλη μπορούν να αναπτυχθούν ταχαίως επειδή βρίσκονται τώρα σε σε φάση ύφεση, αυτή η εξοικονόμηση ενέργεια ω υποχρέωση αποτελεί κίνδυνο για την ανάπτυξη αυτή. Γι' αυτό Θέλουμε να υπάρξει ένας δείκτης εξοικονόμησης της ενέργειας όπου θα υπάρχουν μέρη ε, μιας ενεργειακής εισρωής και να μπορεί αυτή να μετρείται ε, σε σχέση με την ανάπτυξη. Ο κύριος Τούρμες σας μην ανησυχεί. Δεν θα αποδυναμώσουμε αυτό που λέει για 368 εκατομμύρια τόνους ε, αερίων. Άλλωστε δεν είναι η μοναδική, ο μοναδικός τρόπος αυτός η οδηγία Νομίζω ότι πλανόμεθα όταν λέμε ότι μόνο με την οδηγία αυτή μπορούμε να επιτύχουμε το 368. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι δρόμοι που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα και α τα προσθέσουμε αυτά όλα και τότε νομίζω ότι καταλήγουμε εύκολα στο στόχο αυτό. Για το 4 και 5 τώρα βέβαια ο δημόσιος τομέας πρέπει να αποτελέσει πρότυπο αλλά θα επιβάλλουμε στις ε, τοπικές κοινότητες να ε, περνούν από εξυγίανση, από άποψη δηλαδή όλα τα κτίρια του σε βαθμό 3% κάθε χρόνο, αυτό ξεπερνά τι οικονομικέ δυνατότητε ε, των ε, τοπικών κοινοτήτων. Εμεί στο Ομοσπονδιακό Κρατήριο του Βραδεμβούργου εξετάσαμε το ενδεχόμενο αυτό και το κόστο εξυγίανση από την οδηγία αυτή ξεπερνούν όλες τις δαπάνες για την ε, κατασκευή δρόμων, ακινήτων κλπ. Μόνο και μόνο αυτή η επιβολή υποχρέωσης. Και σιγά σιγά αυτά, αυτές οι υποχρεώσεις ανταγωνίζονται ουσιώδεις δαπάνες των ε, τοπικών ε, κοινοτήτων για άλλα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι σημαντικό βέβαια το θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα στο το επίπεδο των τοπικών αυτοδιοίκησεων. Το άρθρο 6 1,5% των, του κύκλου εργασιών μείωση. Μπορούμε τώρα να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις υπεύθυνε για την δράση των πελατών τους. Είναι σοβαρό αυτό. Δεν βγάζουμε έτσι έξω τις μικρές βιοτεχνίες όταν πλέον οι μεγάλοι προμηθευτές ενέργειας έρχονται και προσφέρουν ενέργεια στα νοικοκυριά. Δεν ανακατεύουμε εδώ τα επίπεδα. Πρόκειται δηλαδή για πράγματα τα οποία μένει ακόμη να ξεκαθαριστούν και διερωτώμεθα εάν δεν θα πρέπει να δοθούν καλύτερα οι δυνατότητε στι χώρε μέλη για να επιτύχουν το μεγάλο στόχο του 20% με λιγότερη γραφειοκρατία, μάλιστα ίσω να επιτευχθεί και νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει και το άρθρο 8, το οποίο έρχεται σε αντίφαση με το τρίτο πακέτο της ενιαίας αγοράς για το roll-out των ευφυών μετρητών που οι χώρε μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν στη βάση μελετών που θα κάνουν και αυτό το λέει και μέσα στο τρίτο πακέτο της ενιαίας αγορά, να προχωρήσουν μετά σε διαπραγματεύσεις και αυτό εδώ έρχεται σε αντίφαση με αυτό που λέμε. Τελευταία παρατήρηση για το άρθρο 10 για την συμπαραγωγή ενέργειας και θερμικής ενέργειας και για την αποθήκευση της ενέργειας. Είναι σωστές οι παρατηρήσεις του κ. Τούρμες αλλά οφείλουν να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Και δεν ξέρω αν αυτή την παρέμβασή μας στο σχεδιασμό τους θα τη δεχθούν οι χώρες μέλη. Το ίδιο πρέπει να είναι δεδομένη η αποδοτικότητα των επενδύσεων αυτών. Όταν έχουμε όπως στη Γερμανία 200 250.000 σχέδια στο κοινοτικό επίπεδο για ε, την συμπαραγωγή αυτή πώς θα τα επεξεργαστούμε και θέλουμε άλλωστε νέα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από ε, φυσικό αέριο, πώς θα συνδυαστεί η προσπάθεια αυτή τώρα με αυτά τα δεδομένα. Εάν απορρίπτονται αυστηρά όλες οι εξαιρέσεις στη βάση των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων. Εν τέλει, η αύξηση της αποδοτικότητας της ενέργειας είναι σωστός στόχος, όμως θέλουμε άλλο ορισμό της αποδοτικότητας της ενέργειας έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσει, να μην τεθεί σε κίνδυνο μάλλον και η ανάπτυξη στις ε, διάφορες χώρες. Θέλουμε να διατηρηθεί η διεπίπεδη προσέγγιση, θέλουμε πρώτα να αναλυθούν δηλαδή επιπτώσεις των μέτρων μας για να είναι εξασφαλισμένη η ε, επιτυχία τους και μετά να τις υποβάλουμε στις χώρες μέλη. Και τρίτο, πρέπει να επιτρέψουμε στις χώρες μέλη περισσότερη ελευθερία και για ε, τις αποφάσεις που θα λάβουν και για το 3% της, ανα, της ανανέωσης εξυγένσης επιβαρύνει υπερβολικά τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Βεβαίως η αποδοτικότητα της ενέργειας έχει πραγματικό νόημα όταν αποδίδει και οικονομικά. Ευχαριστώ. Ερτσόκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σκιώδη συζητήτριά μας δεν είναι παρούσα σήμερα και μου ζήτησε να μεταφέρω σε ένα σημεία για την οδηγία αυτή ε, και απλά θα σας τα μεταφέρω. Λέγει ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο μήνυμα το οποίο θα στείλει το Κοινοβούλιο προς το Συμβούλιο. Το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίζει την εικόνα την οποία έχουμε εμείς για την, ε, την αποτελεσματικότητά μας στον τομέα της ενέργειας. Το θέμα δεν είναι να πούμε ναι θα είμαστε αποτελεσματικοί ή δεν θα είμαστε. Το θέμα είναι να στραφούμε στο μέλλον. Θα πρέπει μόνο εφόσον στραφούμε στο μέλλον να αποκτήσουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα της αγοράς της ενέργειας. Το θέμα του κόστους της ενέργειας ε, συνολικά είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Αν δει κανεί τι εξελίξεις των τιμών του πετρελαίου τα τελευταία 10 χρόνια, θα δει ότι η πραγματική τιμή στην ουσία λίγο έχει ξεπεράσει την τιμή στην οποία είχε φτάσει τη δεκαετία του 70 μετά από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο την ενέργεια είναι σε θέση να κάνουν πραγματική εξοικονόμηση κόστους. Το θέμα δεν είναι μόνο η τιμή βέβαια, είναι και η ασφάλεια. Η χρήση ακριβώς αυτών των καυσίμων δημιουργεί εξαρτήσεις. Είμαστε εξαρτημένοι από πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις διακοπής προμήθειας Είμαστε εκτεθειμένοι με λίγια λόγια στην αγορά αυτή της ενέργειας, κάτι το οποίο θίγει τις οικονομίες μας. Και τέλος υπάρχει φυσικά πολύ σημαντικό και το θέμα του ενεργειακού ίχνους. Το ίχνος μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ε, παραγωγής ε, διοξιδίου του άνθρακα είναι αυτό το οποίο είναι πρέπει να θέσουμε δεσμευτικούς στόχους στον τομέα της αποτελεσματικότητας λοιπόν της χρήσης της ενέργειας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία εναλλακτική δυνατότητα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ενεργειακή μας πολιτική θα πρέπει να είναι επίσης και μια δίκαιη πολιτική πάρα πολλοί κόσμος στην Ευρώπη ξοδεύει πάρα πολλά χρώματα, χρήματα συγγνώμη, για την ενέργεια, για την προμήθεια ενέργειας. Αυτό δημιουργεί κοινωνικές αδικίες. Τα άρθρα 6 και 12 αναφέρονται στις κοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα προγράμματα ενεργειακής αποτελεσματικότητας και η Ρίκα Τόμψεν προσπαθεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις διατυπώσεις αυτές. Πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσω εκ μέρους της Μπρίτα για τις προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει και πράγματι η οδηγία αυτή είναι πολύ φιλόδοξη και πολύ σωστά. Ευχαριστώ λοιπόν εκ μέρους της Μπρίτα. Ευχαριστώ. Ρόντε παρακαλώ. Είμαι και εγώ αναπληρωτής. Ίσως μπορούμε να τα καταφέρουμε σε σχέση με το την ιδιότητά μας ως ε, αναπληρωτών. Εν πάση περιπτώσει κύριε Τούρμες, το έργο αυτό για την έκθεσή σας ε, έρχεται σε μια χρονική στιγμή που είναι σημαντική, όπου η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα μπορούσε να έχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με καινοτομία, δημιουργώντας τοπικές θέσεις απασχόλησης, προωθώντας την οικονομία και εξοικονομώντας κονδύλια στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις και στις δημόσιες αρχές οι στόχοι δίνουν αποτελέσματα όπως δίνουν ένα πλαίσιο επενδυτικής ασφάλειας για τη βιομηχανία και δείχνουν ότι υπάρχει και πολιτική δέσμευση να είμαστε αποτελεσματικοί. Επιπλέον οι εθνικοί αποδοτικοί στόχοι για την ενέργεια ευθυγραμμίζονται με την ατζέντα και την αρχή της επικουρικότητας. Έτσι αποφεύγουμε ε, υπερβολικά δεσμευτικά μέτρα σε σχέση με τα κράτη-μέλη και έχουν ένα ευλίγιστο πλαίσιο τα κράτη-μέλη για να είναι αποτελεσματικά και να εξοικονομούν ενέργεια όσον αφορά τις εθνικές τους ανάγκες. Καλωσορίζουμε την προσέγγιση του εισήγητη να επικεντρωθεί <clears throat> στα χειρότερα όσον αφορά την αποδοτικότητα δημόσια κτίρια, κρατικά κτίρια και από πλευράς της ε, συμπληρωματική προσέγγιση όσον αφορά την οδηγία για τα κτίρια ε, του 2010 θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί όσον αφορά το νομικό πλαίσιο. Όσον αφορά τα κτίρια, τελικός μας στόχος είναι να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Θα ήταν χρήσιμο τα κράτη-μέλη να υπολογίσουν το ποσοστό της μείωσης όσον αφορά τους στόχους, όσον αφορά την κατανάλωση σε σχέση με τα κρατικά κτίρια αυτό επίσης θα έδινε πάλι μεγαλύτερη ευληγησία στις κρατικές αρχές. Πώς θα μπορούσαν να μειώσουν την κατανάλωση ενεργειακών πόρων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την υποχρέωση όσον αφορά την ε, κάλυψη των ενεργειακών ε, ε, αναγκών. Είναι σημαντικό να είμαστε φιλόδοξοι, να διατηρηθεί ο στόχος του 1,5% όμως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευλήγησία πώς θα το πετύχουν αυτό δεδομένης της πολυμορφίας μηχανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη. Ο εισηγητής έχει εισαγάγει κάποιες καλές βελτιώσεις για το άρθρο 8 όσον αφορά και την παρακολούθηση αυτή. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι καταναλωτές την κατανάλωσή τους ε, την δυνατότητα εξοικονόμησης όσον αφορά τις υπηρεσίες που τους παρέχονται και πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός όσον αφορά ένα λογαριασμό για την ε, ε, κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών που πρέπει να εξοφληθεί και ένα λογαριασμό σε σχέση με καταλεπτόσα που θα αντανακλά την κατανάλωση ενέργειας από πλευρά των καταναλωτών. Σε σχέση με τα μέτρα που προτείνονται σε αυτή την οδηγία όσον αφορά αφορά την θα πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα τα οποία προτείνονται για την ζήτηση από την άλλη πλευρά όσον αφορά ιδιαίτερα την οδηγία για τα κτίρια Καλοχαιρετίζουμε τα νέα εδάφια από πλευρά εισηγητού στο άρθρο 12, την ανταπόκριση στην ζήτηση. Αυτή η ανταπόκριση στη ζήτηση πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως και άλλα μέσα σε σχέση με την κατανάλωση σε χρόνους εχμής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οι ενεργειακές αγορές να ευθυγραμμίζονται. Αυτά είναι όλα όσα είχα να πω ε, ζητώ συγγνώμη για τις δυσκολίες ίσως ε, που προκάλεσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κάριν παρακαλώ. Well, with the Λοιπόν, σύμφωνα με την παράδοση την οποία φαίνεται ότι δημιουργούμε και εγώ αναλαμβάνω σήμερα το ρόλο να παίξω την κυρία Βίκη Φόρντ. Όλοι κάποιος άλλος είμαστε. Δεν μπορεί να είναι παρούσα η κυρία Φόρντ, αλλά μου ζήτησε να σας διαβάσω την εξής στήλωση. Γι' αυτό λοιπόν θα σας τα διαβάσω λίγο μονότονα, ε, αντίθετα από αυτά τα οποία έκανε ο συνάδελφος πριν. Η Βίκη θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την προσπάθεια που έκανε, υποστηρίζει τους στόχους της οδηγίας, αλλά θεωρεί η Βίκη ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν αρκετή ευελιξία για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Όπως υπόθηκε και στην τελευταία συζήτηση, θα ήθελε το θέμα της οδηγίας για την αποτελεσματικότητα της ενέργειας να υποστηριχθεί από το σύνολο των κρατών μελών και όχι να μπούμε σε διαπραγματεύσεις εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εναντίον του Συμβουλίου. Θα καταθέσει η Βίκη τροπολογίες για τα δημόσια κτίρια γιατί αν υπάρξει αναγκαστική συμμόρφωση σε αυτή την περίπτωση δεν θα αλλάξουν οι στάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτηρίων. Σχετικά με το άρθρο 5 πρέπει να ενισχύσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες να μεγιστοποιήσουν ε, με τον τρόπο λειτουργία τους την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Όχι, ε, να, όχι παρεμβαίνουμε ε, ατομικά Σχετικά με το 6, στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ενέργειας, όχι η μείωση στην κατανάλωση. Θα ήθελα τα κράτη-μέλη να έχουν περισσότερους στόχους για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν ένα επιπλέον κόστος σε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή το συγκεκριμένο εξοπλισμό δεν συμφωνεί με την κατάργηση των εξαιρέσεων του άρθρου 10 που προτείνει ο εισηγητής. Θεωρείται το σύνολο του άρθρου αυτού, το οποίο είναι περιοριστικό και ε, δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με την πιθανή χρήση άλλων μορφών ενέργειας όπως οι εναλλακτικέ και η πυρηνική ενέργεια στο μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να εξαιρέσουμε και τις μονάδες της πυρηνικές από την υποβολή τους σε συγκεκριμένες τεχνολογικές απαιτήσει. Θα πρέπει να πω ότι η Δίκη θα προχωρήσει σε μια προσπάθεια να βρεθούν συμβιβασμοί σε συνεργασία με τον εισηγητή έτσι ώστε να υπάρξει ενεργειακή αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη, από τις βέλτιστες πρακτικές οι διάφορες χώρες να ωφεληθούν, διατηρώντας την εύρυθμη λειτουργία των αγορών στο σύνολο της Ευρώπης. Και τώρα επιστρέφω στο ρόλο μου ως κύριος Καρίμ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αν στο μέλλον ε, συμβαίνει πιο συχνά αυτό, ας γίνεται καλύτερα ανταλλαγή επιστολών. Δεν χρειάζεται να συναντώμεθα. Βέβαια, η πολιτική συζήτηση συνίσταται στην ανταλλαγή επιχειρημάτων και ίσως θα πρέπει να γίνει πια με άλλον τρόπο αυτή η ανταλλαγή επιχειρηματία, ότι αλλιώς δεν έχει καθένας παρά να πει την άποψή του και να βάλει μια τελεία μετά. Τώρα ο συνάδελφος Βιδάλ Κουάδρας λαμβάνει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω για το άτομό μου εγώ προσωπικά. Εντάξει παρεμβαίνω. Ε, Σήμερα έχουμε μια πρώτη, ένα πρώτο γύρο συζήτησης ε, χαρακτήρα, ας το πω έτσι, εκ προημίου συζήτηση. Αυτή η οδηγία θα έχει πολλά θέματα που θα καλύπτει, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα ότι ο φίλος μας Κλοντ Τούρμες κατέθεσε 119 τροπολογίες. Έτσι λοιπόν θα έχουμε πολλή δουλειά στο μέλλον σίγουρα. Το πρώτο που θα ήθελα να επισημάνω, Πρόεδρε, είναι ότι τα θεμέλια από πλευράς προσέγγισης αυτής της οδηγίας, τα θεμέλια πρέπει να είναι σαφή και υπάρχουν δύο δυνατότητες προσέγγισης από πλευράς φιλοσοφίας που δεν συμπίπτουν οι δύο. Στη μία τίνεται, ε, υπογραμμίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας όσον αφορά απόλυτους όρους, δηλαδή μείωση της κατανάλωσης σε απόλυτους όρους. Και η άλλη γραμμή προσέγγισης ως φιλοσοφία είναι, τονίζει, τη δράση στη βελτίωση της αποδοτικότητας, ενεργειακής αποδοτικότητας. Με άλλα λόγια, την ενέργεια που καταναλώνουμε πρέπει να έχει μεγάλη αποδοτικότητα. Αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά ότι είναι εκείνο που πρέπει να αναζητήσουμε, να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα στον ενεργειακό τομέα. Δηλαδή κάθε φορά να κάνουμε περισσότερα, καταναλώνοντας λιγότερα, λιγότερα καύσιμα. Διότι αν έχουμε αιμονή απλά με την μείωση σε απόλυτους όρους, μπορούμε να φτάσουμε στο παράδοξο στο ότι θα καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια και θα είμαστε λιγότερο αποδοτικοί. Πράγμα το οποίο θα ήταν δραματικό και παράλογο. Υπάρχει μια δυναμική των πραγμάτων λοιπόν όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη στις προηγμένες ε, οικονομίες του κόσμου. Υπάρχει ένας τρόπος ε, δημιουργίας ε, πλούτου και απασχόλησης και που πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα υποχρεωτικά ότι πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να είμαστε κάθε φορά πιο αποδοτικοί, πιο αποτελεσματικοί. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, πολλά άλλα πράγματα θα είναι πιο εύκολα και θα διευκολυνθούν και θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επ' αυτών. Και παρέμεινα ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο διότι είναι τα, τα θεμέλια τα βάθρα όλης της συζήτησης που πρέπει σε αυτά να βασιστούμε. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε ένα σημείο σύγκλησης και συμφωνίας. Μετά, όσον αφορά το άρθρο 6. Στο άρθρο 6 θεσπίζεται ένα καθεστώς υποχρεώσεων εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά τις ενεργειακές επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας. Στο ίδιο αυτό άρθρο ομολογείται επίσης ότι μπορούν να υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα. Όμως μόνο αν αυτά τα εναλλακτικά μέτρα εγκρίνονται, έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, α τα πάρουμε ένα προ ένα. Μία συμμετρική σχέση υπάρχει εδώ που δεν θεωρώ ότι είναι η πιο, η πιο ορθή. Και τα δύο πράγματα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο και να αντιστοιχούν. Και η εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων αλλά και τα εναλλακτικά μέτρα στο ίδιο επίπεδο θα πρέπει να μπορούν να, προχωρήσουν αν υπάρχει προηγούμενη έγκριση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλο πράγμα είναι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βλέπει στη συνέχεια αν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις που έχουν επομιστεί τα κράτη-μέλη αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε, να εισαγάγουμε μια αρνητική διακριτική μεταχείριση σε σχέση με αυτές τις δύο εναλλακτικέ δυνατότητες να αναζητηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα, υλοποιώντας πάντα τους στόχους, συμμορφούμενοι προς τους στόχους. Και εν τέλει, τελευταίο, θα ήθελα να αναφερθώ σε σχέση με τη συμπαραγωγή ενέργειας και θερμότητας. Η συμπαραγωγή ενέργειας θερμότητας όχι μόνο είναι η παραγωγή θερμότητας, ε, δυνατότητας ε, κατάψυξη, ε, Υπάρχουν βιομηχανίε με άλλα λόγια που χρησιμοποιούν τη συμπαραγωγή ως μέρος, τμήμα της παραγωγικής δυνατότητάς τους, ως του προτύπου παραγωγικής δυνατότητας. Διότι έτσι έχουν την καλύτερη αντιμετώπιση των πόρων και είναι πιο αποτελεσματικές. Γι' αυτό α διευρύνουμε τον οριζοντά μα το φάσμα αυτό και να ξέρουμε ότι η συμπαραγωγή της ε, ψήξης και της ε, θέρμανσης μαζί με την παραγωγή ενέργειας και πολλά άλλα πράγματα είναι παραγωγικά σε σχέση με το βορρά της Ευρώπης και το νότο της Ευρώπης που έχουν ιδιομορφίες. Με αυτό τον ευρύτερο ορίζοντα είναι προφανές πλέον ότι η συμπαραγωγή Καμιά φορά είναι σκόπιμη, καμιά φορά όμως δεν είναι η πιο αποτελεσματική. Δεν μπορούμε να θεσπίσουμε καθολική οικουμενική υποχρέωση να υπάρχει συμπαραγωγή πάντα και παντού, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη σκοπιμότητα και την κερδοφορία και τις ιδιομορφίες που εξαρτούνται όχι μόνο από την ανάγκη να υπάρχει θερμότητα, παραγωγής θερμότητας, αλλά και από πολλά άλλα πράγματα. Μεταφορά καυσίμου, διαδικτύωση, δυνατότητα πρόσβαση στα δίκτυα, κόστος και πολλούς άλλους παράγοντες που πρέπει να σεβόμαστε σκεφτόμαστε και να λαμβάνουμε υπόψη. Γι' αυτό αν οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής μόνο συνδέονται με ένα παράγοντα μπορούμε να καταλήξουμε σε παράλογες καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ πάλι πρέπει να προσαρμόσουμε το όραμά μας στο πιο αποτελεσματικό. Όσον αφορά τη συμβατότητα συμπαραγωγής με άλλες πηγές ενέργειας, να τα πάρουμε πάλι ένα προς ένα. Υπάρχουν πρότυπα σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που απαιτούν οι ενεργητικοί πόροι που θα χρησιμοποιούνται να είναι της μιας μορφής ή της άλλης. Και αυτό έχει επιρροή, επηρεάζει την συμπαραγωγή. Υπάρχουν συμπαραγωγές που απαιτούν λειτουργία της εγκατάστασης 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα πάντα. Ενώ άλλες ε, σε σχέση με την ε, ε, ηλιακή ενέργεια έχουν διαφορετική λειτουργία. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε σχέση με τις ενεργειακές πηγές, για παράδειγμα στα ανανεώσιμα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την βιομηχανική συμπαραγωγή που δεν θα ήταν ίσως η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος η ηλιακή για αυτή τη συμπαραγωγή. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες λοιπόν και να μην είμαστε ε, μονοδιάστατοι όσον αφορά την παραγωγή γιατί μπορεί να οδηγηθούμε σε σφάλματα διαφορετικά. Αυτά είναι οι παρατηρήσεις που είχα να κάνω σε σχέση με τις προκαταρκτικές αυτές παρατηρήσεις στη συζήτησή μας. Έχουμε πολλή δουλειά όπως είπα πρόεδρε να κάνουμε. Υπάρχουν πολλά άλλα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν και από άλλους συναδέφους που και αυτά είναι σημαντικά και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και γνωρίζοντας όλα αυτά το τάλαντο και το ανοιχτό πνεύμα του εισηγητή και την κατανόηση που δείχνει ο εισηγητή, είμαι βέβαιος ότι στο τέλος τέλος θα καταλήξουμε σε μια κοινή θέση και συμφωνία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Δυστυχώς δεν είχα προσέξει πριν τον κύριο Προβέρα. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Τούρμες, για την ε, διαθεσιμότητα την οποία επέδειξε να ακούσει και να δώσει προσοχή, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις. Βάση περιπτώσει, οι στόχοι της οδηγίας ε, είναι σωστοί, ευκταίοι, αλλά για να επιτευχθούν θα πρέπει να είναι και εφικτοί Η πρώτη παρατήρηση που κάνω λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις μεγάλες διαφορές οι οποίες υπάρχουν στην Ευρώπη. Είναι διαφορές όχι μόνο κλιματολογικές, γεωγραφικές ή οικονομικές, αλλά και κοινωνικές και γιατί όχι και πολιτιστικές. Αυτές οι διαφορές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αν σκεφτεί κανείς τι συμβαίνει στις βόρειες χώρες σαν παράδειγμα και δούμε τα χαρακτηριστικά τους, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές με τον νότο της Ευρώπης. Η πρόταση λοιπόν του να δημιουργηθεί στην Ευρώπη η τηλεθέρμανση και η από κοινού παραγωγή ε, θέρμανσης είναι κάτι το πάρα πολύ σωστό μεν, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή κατανομή των δημοσίων πόρων, γιατί και εδώ υπάρχουν εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Θα έβλεπα ευνοϊκά το να υπάρξει μια οδηγία η οποία να επιβάλλει συγκεκριμένους στόχους στα κράτη-μέλη, αφήνοντας βέβαια στα κράτη-μέλη την δυνατότητα επιλογής των πλέον αποτελεσματικών και κατάλληλων τρόπων εξοικονόμησης χρημάτων και αποτελεσματικότητας ενεργειακής. Υπάρχουν χώρες που έχουν επιβάλει μέτρα εξοικονόμησης και χώρες οι οποίες δεν έχουν κάνει αυτά τα οποία θα οφείλαν. Σχετικά με τα δημόσια ελλείμματα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε και τη διοικητική και την οικονομική δυνατότητα των κρατών μελών σε σχέση με το 3%. Υπάρχουν ορισμένα ιστορικά κτίρια στις διάφορες χώρες αρχιτεκτονικής αξίας που θα πρέπει να εξεταστούν ε, ξεχωριστά και να εξαιρεθούν ίσως από την οδηγία. Εμείς στη χώρα μου έχουμε σημαντικά προβλήματα οικονομικά αλλά έχουμε και πάρα πολλά διοικητικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους Δήμους να δαπανίσουν τους πόρους που ήδη έχουν στη διάθεσή τους και έχουμε και μια περίεργη κατάσταση πολλών ιστορικών κτηρίων αρχιτεκτονικής αξίας που χρησιμοποιούνται από το κοινό για διάφορους στόχους. Ένα άλλο θέμα είναι να συνδυάσουμε την ενεργειακή αποτελεσματικότητα με την πολύ ευκταία οικονομική ανάκαμψη. Πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας λοιπόν στην αποτελεσματικότητα και όχι τόσο στην εξοικονόμηση να δούμε το θέμα της αποτελεσματικότητας ε, με φιλόδοξο τρόπο γιατί πολλές φορές κάποιες υπερφιλόδοξες οικολογικές τάσεις δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία. Θα συμφωνήσω και με τον εισηγητή όταν λέει ότι πρέπει να βρεθούν και τα ε, χρηματοπιστωτικά μέσα ε, για να, γιατί αλλιώς στην ουσία θεωρητικολογούμε. Είναι η αλήθεια ότι εδώ θα πρέπει να βοηθήσουμε την ε, δυνατότητα ανάπτυξης της βιομηχανίας η οποία θα πρέπει να ανοίξει σε νέες τεχνολογίες, νέες έρευνες, να υπάρξει έστω και μια νέα μορφή οικονομικής ανάκαμψης. Σημασία έχει επίσης και η ενημέρωση των πολιτών. Πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες ε, τι ακριβώς συμβαίνει ε, μέσα από την ευαισθητοποίηση των πολιτών θα πρέπει να τους πείσουμε να χρησιμοποιήσουν καλύτερα την ενέργεια που έχουν στη διάθεσή τους και να αποκτήσουν φυσικά μια νέα αντίληψη πράσινη οικολογική την οποία ο κύριος Τούρμες σίγουρα θα υιοθετήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μπέλετ. Ευχαριστώ. Λίγα σχόλια στα Ολλανδικά, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας μέχρι τώρα. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ορισμένα από τα όσα ήθελα να πω ήδη καλύφθηκαν και θα τα επαναλάβω. Για παράδειγμα, για το κριτήριο του εμβαδού ανατετραγωνικά. Και εκεί πιθανόν το κριτήριο αυτό να μην είναι το καλύτερο και ίσως είναι καλύτερα να ε, είναι το κριτήριο η συνολική ε, κατανάλωση του ε, κτηρίου. Ίσως λοιπόν το κριτήριο των τετραγωνικών να πρέπει να επανεξεταστεί. Δεύτερο τώρα, οι αναθέσεις δημοσίων έργων, δημόσιες αναθέσεις και ούτε καθεξής. Βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη εδώ ότι πάντοτε επιλέγεται ο φθηνότερος που όμως δεν είναι απαραίτητα και ο ενεργειακά αποδοτικότερος ε, ομοιοδότης δηλαδή. Αυτό πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη. Τρίτο, carbon leakage, διαρροή, δηλαδή εννοείται των επιχειρήσεων για να ε, εγκατασταθούν αλλού. Αυτό δεν επιβαρύνει ιδίω τις ε, πιο ε, τις, ε, τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια και αυτές δηλαδή μετεκαθίστανται, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό στους εθνικούς σχεδιασμούς και το ενδεχόμενο δηλαδή αυτά, να, αυτές να εξεταστούν ιδιαίτερα. Οι επιπτώσεις δηλαδή για τις επιχειρήσεις οι οποίες καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια και ο κίνδυνος να μετεκατασταθούν. Τέλος, οι τελικοί καταναλωτές, οι τελικοί χρήστες της ενέργειας. Απευθύνω έκκληση προς όλες και όλους τους συναδέλφους να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο όταν πρόκειται δηλαδή πλέον για τους λογαριασμούς του ρεύματος διότι στις περισσότερες περιπτώσεις εκεί αναφέρεται μόνο το κόστος της ενέργειας. Χρειάζεται να υπάρξει όμως πολύ περισσότερη διαφάνεια. Όχι μόνο δηλαδή το κόστος της ενέργειας αλλά και το κόστος της διανομής πρέπει να αναφέρεται στους λογαριασμούς αυτούς. Καθώς επίσης και οι υποχρώσεις ε, δημοσίων υπηρεσιών, οι public service obligations των ε, προμηθευτών που έχουν ορισμένες υποχρεώσεις να εκπληρώσουν και αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ιδίω δηλαδή στο άθρο που ε, αναφέρεται στους λογαριασμούς της ενέργειας θέλουμε να υπάρχουν και μεγαλύτερη διαφάνεια και πολύ περισσότερες πληροφόρειες προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Ευχαριστώ κύριε Μπέλετ, η κυρία Κολάνσκα Παπίνσκα. Ο λόγος για τον οποίο λαμβάνουν τον λόγο τα δύο αυτά πρόσωπα, ο κ. Μπέλετ και η κ. Παπίνσκα, είναι ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν μπόρεσαν να μιλήσουν. Πρώτα κυρία Κολάσκα Παπίνσκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω την αγγλική τελικά. Εμείς ε, δεν είχαμε ρυθμίσει το θέμα αυτό και το περιμέναμε την πρόταση εδώ και αρκετό καιρό. Θα επηρεάσει και την οικονομία και τις τοπικές αρχές, τις τοπικές διοικήσεις, ε, το δημόσιο και τα νοικοκυριά. Οι επιπτώσεις οικονομικά θα είναι διαφορετικές και θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Μιλώντας για την οικονομία, είναι κρίσιμη η σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ενεργειακή ε, αποδοτικότητα. Η ενεργειακή αποδοτικότητα σημαίνει μια μετακίνηση προς εξοικονόμηση ενέργειας γενικότερα, ιδιαίτερα για τις οικονομίες οι οποίες αναπτύσσονται με αργότερους ρυθμούς θα πρέπει αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας στους κανονισμούς τους οποίους ε, θα ψηφίσουμε. Οι αλλαγές σε οικονομίες ε, της ε, Δανίας ή της Σλοβακίας θα επηρεάσουν διαφορετικά γενικότερα την κατάσταση στις χώρες αυτές και τα δημοσιονομικά τους. Συμφωνώ με αυτούς που λέγουν λοιπόν ότι ε, θα πρέπει αναμονάδα να αντιμετωπίζεται η αποδοτικότητα και όχι σε απόλυτους αριθμούς. Γιατί οι αναπτυσσόμενες οικονομίες πρέπει να μην εμποδιστούν να χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια. Πρέπει να τη χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά, αλλά δεν μπορούμε να τους ζητάμε να αυξάνουν τους φόρους με τέτοιο τρόπο. και δεν πρέπει να υποστηρίζουμε τις χώρες αυτές συστηματικά με χρήματα που προέρχονται από άλλες χώρες μέσω του Περιφερειακού Ταμείου. Τώρα η απέτηση 3%. από τις περιφέρειες και από τις τοπικές αρχές. Νομίζω ότι έχει σημασία καταρχάς να θέσουμε στόχους πολιετής, όχι ετήσιους αυστηρά για τις ορισμένες περιπτώσεις ε, τα κρατή μπορεί να ξοδεύουν περισσότερο και άλλες χρονιές λιγότερο. Ας μην αποφασίσουμε λοιπόν σε ένα 3% αλλά ας δούμε λίγο πιο μακριά. Το ίδιο αφορά επίσης και τους ελέγχους ε, για την ενέργεια, τις ελεγκτικές διαδικασίες. Νομίζω κάθε δύο χρόνια είναι υπερβολικό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μερικές φορές γρήγορα, μερικές φορές αργά και υπάρχουν διαφορετικές ε, ταχύτητες στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Κάποιες από τις ε, κοινωνίες, τις τοπικές, ε, θα θεωρήσουν ότι το 3% είναι υπερβολικό και ζούμε επίσης και σε μία περίοδο κρίσης κυβερνήσεις ε, περνούν δαπάνες ε, για, ε, για το δικό δίκτυο, για τα σχολεία, για την υγεία και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και πολλές τοπικές τέτοιες αρχές έχουν τεράστια ελλείμματα και θέλουν να, κάνουν εξοικονομήσεις μειώνοντας τον δημόσιο φωτισμό σαν παράδειγμα. Αλλά δεν πρέπει να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα των προμηθειών. Σε ορισμένε ε, περιοχές, λιγότερο αναπτυγμένες, πιο γεωργικές αν θέλετε, αν μου ζητήσουν να επιλέξω πιο αποτελεσματικά μέσα και προϊόντα, θα επιλέξω τα προϊόντα τα οποία ίσως μερικές φορές να παράγονται μακράν σε άλλες χώρες, γιατί δεν υπάρχουν τοπικά προϊόντα αντίστοιχα που θα μπορούσαν να επιλεγούν. Αυτό ισχύει σαν παράδειγμα για αυτούς οι οποίοι παράγουν κουφώματα ή παράθυρα στις διάφορες χώρες. Λοιπόν, το πιο αποδοτικό ενεργειακά είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα τις τοπικές συνθήκες και ένας από τους συναδέλφους αναφέρθηκε και στο θέμα της σωστής ενημέρωσης και δεν πρέπει να μην το περιλάβουμε αν θέλουμε να γίνουν αλλαγές στην οικονομία και στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας των κοινωνιών μας θα πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στην ενημέρωση και δεν θα πρέπει το θέμα αυτό να αφορά μόνο τους πολιτικούς αλλά να υπάρξει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή εκστρατεία γύρω από την ενημέρωση για αυτό το τομέα. Η κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μάλιστα, ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Σημαντικό και είναι το για ποιον κάνω λόγο εγώ, εξ ονόματος τίνος ομιλώ, εξ ονόματος των μικροπαραγωγών ενέργειας, εκείνοι που θα ήθελαν να παράγουν ενέργεια στα νοικοκυριά τους για παράδειγμα, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες αυτών των νοικοκυριών, σε σχέση με εκείνους που εισέπραταν από πλευράς μεγάλης παραγωγής τέλη και σε σχέση με την αποδοτικότητα. Είναι όμως σημαντικό την άλλη πλευρά ήδη οι νοικοκύριδες να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη στα νοικοκυριά τους για αυτού του είδους την παραγωγή. Πολλά νοικοκυριά στην χώρα μου, την Ολλανδία, βρίσκονται στα χέρια ε, τέτοιων ε, δυνατοτήτων, ας το πω έτσι, από πλευράς παραγωγής και θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα παραγωγής από πλευράς τους. Αυτό θα σήμαινε ότι ένας νοικοκύρης θα είχε τη δυνατότητα να είναι έτσι πιο αποτελεσματικός. Ας δώσουμε λοιπόν άδεια και δυνατότητα οι νοικοκύριδες αυτοί, οι ε, κάτοχοι νοικοκυριών να πάρουν την παραγωγή στα χέρια τους. Σημαντικό είναι αυτό. Μικροπαραγωγή είναι κάτι που θέλουμε να προαχθεί. Θέλουμε να εμπλακούν οι πολίτες στην παραγωγή και να έχουν τη δυνατότητα πέρα από την κατανάλωση να μπορούν να παράγουν και οι ίδιοι ε, τέτοιου είδους ε, ενεργειακούς πόρους. Ε, είναι σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρεται από πλευράς συναδέφου, αλλά θα πρέπει να μπορεί να εντάσσεται και να προσαρμόζεται αυτή η πρόταση και σε σχέση με άλλες οδηγίες. Οδηγίες για την κτηριακή αποδοτικότητα όσον αφορά την ενεργειακή χρήση. Και άλλες τέτοιες προτάσεις που βρίσκονται καθοδόν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες μορφές αποδοτικότητας, πέρα από την ενεργειακή αποδοτικότητα και δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε ε, ή να έχουμε μόνο ε, θέματα επισκευών θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά τους λογαριασμούς ε, που καλούνται να εξοφλεί να πληρώσουν ε, οι καταναλωτές. Αυτή η οδηγία αλλά και μελλοντικές οδηγίες προφανώς εγώ ε, εστιάζομαι σε αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία πρέπει να δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να είναι αποτελεσματικοί. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια σαφή εικόνα για την κατανάλωση ενέργειας και τους λογαριασμούς που τους αποστέλλονται. Η πληροφόρηση είναι πάρα πολύ σημαντική και ξεκινά όσον αφορά την πληροφόρηση για την κατανάλωση Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια οργανωτική, αν θέλετε, διοργανωτική παρατήρηση. Αναβλήθηκε η κίνηση, τα εγγένεια του Γαλιλαίου. Δεν θα γίνουν σήμερα, αλλά αύριο. Είχα υπόψη μου ότι θα είχαμε χρόνο, αλλά ήταν μια μικρή ελπίδα αυτή. Διότι οι διερμηνείς είναι πρόθυμοι να μας δώσουν μόνο ένα τέταρτο, αλλά όχι παραπάνω. Αλλά μπορούμε να δραχθούμε τι ευκαιρίες να εκμεταλλευτούμε αυτά τα 15 λεπτά. Έχω 5 συν τον Κλοντ, συν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητούν να παρέμβουν. Παράκλησή μου να προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι ώστε όλοι να παρέμβουν. Η κυρία Τικάου είναι η επόμενη. Παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη μπορώ. Τα μέτρα τα οποία συνδέονται με την αποδετικότητα στον τομέα της ενέργειας ε, έχουν μεγάλο βάρος. Πρόκειται για τον πιο φθηνό τρόπο να εξοικονομήσουμε ενέργεια στο μέλλον. Αυτό το 3% τώρα. και τα μέτρα γενικότερα που προτείνονται για, την αναγκαστική, ε, για τον αναγκαστικό εξυγχρονισμό των δημοσίων κτηρίων. Το 3% της επιφάνειας είναι ένα στόχος πολύ δεσμευτικός. Σαν εισηγήτρια της οδηγίας που αφορά την ενεργειακή αποδετικότητα των δημοσίων κτηρίων, είμαι φυσικά υπέρ του συγκεκριμένου στόχου οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα, θα πρέπει να είναι οι πρώτες οι οποίες θα εξυγχρονίσουν το κτίρια τους, αλλά είναι πάρα πολύ δεσμευτικό και δίσκαμπτο το μέτρο αυτό και νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει την βελτίωση στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία, να έχουν περισσότερες δυνατότητες οι μηχανισμοί και να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την ενεργειακή αποδοτικότητα χωρίς να αναφερόμεθα σε συγκεκριμένα ποσοστά τετραγωνικών μέτρων. Τώρα για τις περιφέρειες. Μία πρόσφατη έκθεση αναφερόταν στο ότι οι αγροτικές περιοχές, η Ήπεθρος, είχε διαφορετικές ανάγκες στον τομέα της προμήθειας ενέργειας από κάποιες άλλες περιφέρειες διαφορετικής φύσεως. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιφερειών, των αγροτικών περιφερειών. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Μπρεζίνα, παρακαλώ. Thank you, Chairman. Uh, some uh, remarks in Czech. Θα τα πω στα τσεχικά, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Κοβάτς για συγγνώμη τον εισηγητή κύριο Τούρμες ήθελα να πω, γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας είναι από τους σημαντικότερους στόχους, στόχους μας. Στην πρόταση ωστόσο που μας έχει υποβληθεί δεν μου αρέσει μια σύγχυση σχετικά με τους ορισμούς της ενεργειακής αποδοτικότητας. Επίσης ε, δεν με ικανοποιεί το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ότι αν δεν επιτύχουμε να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή αποδυτικότητα, αυτό δεν σημαίνει Νομίζω ότι δεν θα, ε, δεν θα μας εξυπηρετήσει. Τι το 1,5% της μείωσης της ε, κατανάλωσης και το 3% των εξοικονομήσεων με την μόνωση, με τη θερμική μόνωση των ε, δημοσίων κτηρίων μου θυμίζουν λίγο λύσεις του παρελθόντος στη χώρα μου. Εάν κανείς είναι σε θέση να επηρεάσουν την ε, συμπεριφορά των καταναλωτών να μειώσουν δηλαδή την κατανάλωση κατά 1,5% εταιρικοί καταναλωτές. Αυτό βέβαια το κατανοώ. Αλλά στην πράξη γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Διότι με την αγοραστική δύναμη του Τσέχου καταναλωτού, για παράδειγμα, η, στην αγοραστική δύναμη μάλλον, η, η το κόστος της ενέργειας είναι μεγαλύτερο, το ποσοστό της ενέργειας, η αναλογία της ενέργειας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες δυτικές χώρες. Εάν λοιπόν είναι έτσι, δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε αυτά με τόσο διοικητικό τρόπο. Για ένα άλλο πράγμα τώρα, που είναι οι διαρθρώσεις της οικονομίας. Σε μια βιομηχανική χώρα έχουμε άλλη κατανάλωση βεβαίως από άλλες χώρες και δεν είναι τόσο εύκολο να αυξηθεί η ανάπτυξη διατηρώντας τα ίδια επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας. Γι' αυτό τα μέτρα αυτά πρέπει να επαναξεταστούν σε βάθος. Δεν θα ήταν καλό στα πλαίσια ενός οράματος μιας πράσινης ε, βιομηχανίας, οικονομίας, να καταστρέψουμε την οικονομία που μας τρέφει τώρα. Κυρία ναι πρόεδρε, να τα πάρουμε ένα προς ένα. Κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων εβδομάδων είχαμε μια σειρά συναντήσεων, ακροάσεων και συναντήσεων συνεδριάσεων άλλου είδους από κάθε πολιτική ομάδα που διοργανώθηκαν. Και υπήρξε ένας κοινό παρονομαστής και αυτός ο κοινό παρονομαστής ήταν το ότι δεν πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ενιαία υποχρεωτικά σε όλα τα κράτη-μέλη για να πετύχουμε τους στόχους της ενεργειακής αποδοτικότητας, διότι η κατάσταση λόγω διαφορετικών λόγων και παραγόντων σε κάθε κράτος μέλος η κατάσταση είναι διαφορετική. Υπήρξαν περιπτώσεις επιτυχίας. Είδαμε πως όσον αφορά την μείωση του διοξιδίου του άνθρακα υπήρξε σημαντική μείωση από κάποια κράτη. Όμως να μεταφέρουμε συγκεκριμένη πύρα ή βίωμα από μια χώρα που συγκεκριμένα μέτρα χρησιμοποίησε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα μεταφέρουμε Εκείνοι που το έκαναν στο τέλος είδαν ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι για την κοινή λογική πρέπει να δούμε ότι είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα, ώστε με ένα κλειδί επιτυχίας αυτής της οδηγίας να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ενεργειακής εξοικονόμησης μέσω αποδοτικότητας για 20% μέχρι το 2020 ή σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, έχει ένα κλειδί, ένα ρόλο κλειδιού παίζει η ευελιξία, η ελαστικότητα. Η ελαστικότητα σημαίνει κάθε χώρα να ξέρει ακριβώς ποιο στόχο πρέπει να υλοποιήσει και να πετύχει και γι' αυτό πόσο πρέπει να συνεισφέρει από πλευρά της. Αυτό είναι το burden sharing, ο επιμερισμός των βαρών και γι' αυτό τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να θεσπίσουν και να καθορίσουν με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και παραμέτρους πόσο κάθε χώρα θα πρέπει να συνεισφέρει και ποιος θα είναι ο στόχος για κάθε χώρα ξεχωριστά. Και από αυτή την αφετηρία να υπάρχει ελαστικότητα, ευελιξία στα μέτρα που θα εφαρμόζονται ώστε κάθε χώρα να μπορεί να πετύχει τους στόχους της. Γιατί καλύτερα τα ξέρουν οι κράτη... τα κράτη-μέλη και κανένας δεν τα ξέρει καλύτερα ποια μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν και ποια μέσα πρέπει να, να ε, εφαρμοστούν για την ε, εισαγωγή προτάσεων από, το Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα όσα λέει ο συγητής πρέπει ενδεικτικό χαρακτήρα να έχουν όλα αυτά και όχι δεσμευτικό. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα monitoring, παρακολούθησης ε, εποπτείας με διαφάνεια που θα επιτρέπει να γνωρίζουμε αν κάθε μια από τις χώρες μας σύμφωνα με την δέσμευση που έχουν αναλάβει για την επίτευξη των στόχων τους ενεργειακής εξοικονόμησης μέσω ενεργειακής αποδοτικότητας αν κάθε μια χώρα υλοποιεί τους στόχους αυτούς ή όχι και ενδεχόμενα θα μπορούσε να υπάρχει η απόσυρση ή η πρόταση αξιολόγησης κάποιων μέτρων που θα πρέπει να στοχεύουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Όμως το κλειδί είναι πρώτον οι χώρες να έχουν ένα σαφή στόχο για αυτές, γι' αυτό μόνο τα κράτη-μέλη γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίζονται οι στόχοι για κάθε χώρα με την Επιτροπή από κοινού για τα μέσα μετά που θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν και να υλοποιούν που πρέπει να είναι μέσα ευέλικτα και ελαστικά που θα αποφασίζουν πάλι κάθε ένα από τα κράτη-μέλη ξεχωριστά για να υπάρχει ευελιξία. Αυτή είναι η βάση με την οποία πρέπει να δράσουμε και να λειτουργήσουμε. Αν θέλουμε πέρα από την ενεργειακή αποδοτικότητα να έχουμε και μια αποτελεσματική οδηγία για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφος Κάριντς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά ακούστηκαν ήδη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω μία διαφορά η οποία απασχόλησε αλλά λίγο κάποιους από τους ομίλητες. Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι το ίδιο πράγμα με την ενεργειακή αποτελεσματικό, αποδοτικότητα μπορεί να πετύχει κανείς εξοικονόμηση με διάφορους τρόπους. Η αποδοτικότητα είναι ένας από αυτούς τους τρόπους. Σβήνοντας τα φώτα επίσης είναι άλλος τρόπος. Μπορούμε να πάρουμε απόφαση, να σβήσουμε τα φώτα, να σβήσουμε τον κλιματισμό και τη θεύμανση και θα εξοικονομήσουμε πάρα πολύ ενέργεια, θα είμαστε πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι μετά, αλλά θα έχουμε εξοικονομήσει ενέργεια. σε μια χώρα, αν τυχόν ας πούμε μειωθεί το ΑΕΠ, μειώνει και την ενέργεια που καταναλώνει. Στη δική μου χώρα, σαν παράδειγμα, εξοικονομούμε πάρα πολύ ενέργεια. Δυστυχώς το υποπροϊόν αυτής της μεθόδου είναι η ανεργία. Έχουμε πολύ ψηλή ανεργία, με υψηλό κοινωνικό κόστος, ο κόσμος δεν έχει δουλειά, εν μέσω της αποτελεσματικότητας το να εξοικονομούμε ενέργεια είναι κάτι το, το οποίο ε, μπορεί να βοηθήσει να τους κρατήσουμε τους ανθρώπους στις θέσεις απασχόλησής τους για να μπορέσουν να δουλέψουν χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια. Βλέπουμε τι γίνεται βέβαια σε αυτή την αίθουσα. Να μην αναμειγνύουμε λοιπόν τις διάφορες ε, έννοιες Τώρα τα 368 εκατομμύρια τόνοι τους οποίους θα πρέπει να εξοικονομήσουμε κτλ. Όλα αυτά ε, μπορεί να είναι σημαντικό κέρδος σε επίπεδο αποδοτικότητας. Όχι σβήνοντας τα φώτα, αλλά ε, κάνοντας το ΑΕΠ της κάθε χώρας να λειτουργεί ε, με αποτελεσματικό και αποδοτικό ενεργειακά τρόπο που να μην δημιουργεί προβλήματα στην ε, οικονομική ανάπτυξη. Είναι σαφές ότι σε διαφορετικές χώρες έχουμε διαφορετικά προβλήματα. Έχουμε χώρες πυκνοκατοικημένες, χώρες αραιοκατοικημένες, χώρες με πολύ ζεστά καλοκαίρια, χώρες με πάρα πολύ κρύους χειμώνες και πάει λέγοντας. Η κατανάλωση ενέργειας λοιπόν ε, και η απλή καλύτερη μόνωση ενός κτηρίου κατά 3% δεν θα βοηθήσει πολύ. Κατά πόσον τα κτίρια αυτά είναι πραγματικά αποτελεσματικά, μπορεί κανείς να πετύχει θετικούς στόχους με σοβαρά μέτρα, αλλά και με μέτρα τα οποία μακροπρόθεσμα δεν είναι σοβαρά. Το θέμα δεν θα είναι λοιπόν τι θα γίνει με το 3% αλλά θα πρέπει αναμέτρο να δούμε τι γίνεται σε κάθε χώρα σε σχέση με τα δημόσια κτίρια σαν παράδειγμα και βλέπουμε τι κάνει η αυτοκίνητο βιομηχανία. Όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο ξέρουμε τι καταναλώνει ε, και τι εκπέμπει ε, ανά χιλιόμετρο. Αυτά είναι μέτρα τα οποία μπορούμε να ε, συγκρίνουμε. Στοιχεία τα οποία μπορούμε να συγκρίνουμε ανάμεσα σε διαφορετικές εταιρείες και μοντέλα. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στα κτίρια. Η αναμονάδα ΑΕΠ σαν παράδειγμα τι ενεργειακή αποτελεσματικότητα μπορούμε να πετύχουμε. Δεν ξέρω τι μορφή μπορεί να πάρει μια τέτοια προσπάθεια, αλλά αυτή είναι νομίζω η σωστή κατεύθυνση. Οι προτάσεις σας είναι καλές και συμφωνώ με τους στόχους της οδηγίας σας, αλλά δεν θα πρέπει εμείς να εμείνουμε στο θέμα της εξοικονόμησης. Αυτό είναι ένα απλό μέσο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Αλλά πρέπει να δούμε πραγματικά ποια μέσα έχουμε στη διάθεσή μας Είπαμε ότι η δική μου χώρα εξοικονομεί ενέργεια. Εμείς έχουμε το 1, 1 τρίτο της ενέργειάς μας που προέρχεται από εναλλακτικέ πηγές. Καλύτερα από άλλες χώρες εκτός από τη Σουηδία. Αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα ότι σε σχέση με το ΑΕΠ είμαστε από τις λιγότερο αποτελεσματικές χώρες στον τομέα της ενέργειας. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια και να παράγουμε περισσότερο προϊόν. Ο κύριος Μπαλσίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφός μου Κάριντς περιέγραψε ορθά την κατάσταση. Πρόκειται για την κατάσταση που ισχύει στις βαλτικές χώρες. Βεβαίως έχουμε πολλά προβλήματα. Έχουμε και βαριά κληρονομιά από την σοβιετική εποχή, πολλά κτίρια που θα έπρεπε να εξηγενθούν η διαδικασία αυτή δεν προχωρεί αρκετά γρήγορα. Έχουμε μεγάλους και φιλόδοξους στόχους, έχουμε συζητήσει πολύ πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Κατά τη γνώμη μου, οι στόχοι αυτοί μπορούν να γίνουν στρατηγικοί στόχοι. Πολλοί δηλαδή από τους επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα μιλούν για πολύ απειλητικές εξελίξεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε λαμβάνοντας μέτρα, συγκεκριμένα μέτρα. Γι' αυτό και χαίρομαι για την πρώτη αυτή εκδοχή του εγγράφου του εισηγητού. Βεβαίως και είναι αδύνατον να λυθούν όλα τα προβλήματα με μία μόνο έκθεση. Γι' αυτό τάσομαι υπέρ της ιδέας κάθε χώρα μέλος να θέσει δεσμευτικούς στόχους, να υπάρχει και έλεγχος για το πώς βαίνει η προσπάθεια επίτευξη των στόχων. Άλλωστε, λέχθηκε ήδη ότι έχουμε διαφορετικές καταστάσεις πρέπει να λάβουμε υπόψη από άποψη κλίματο, γεωγραφίας κλπ. Θα πρέπει επίσης να ε, συζητήσουμε και το θέμα των ε, αναθέσεων δημοσίων έργων και να κατανοήσουμε ότι στόχος μας, στόχος δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι η τροποποίηση του καθεστώτος ε, των δημοσίων αναθέσεων στις οποίες ο ανθρώπινος παράγων δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Έτσι θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Το σύστημα έχει ήδη δημιουργηθεί. Είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. Γνωρίζουμε όλοι για ποιο λόγο. Και γι' αυτό υποστηρίζω τις ιδέες του εισηγητού και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Να δώσουμε σύντομα το λόγο στην Κομισιόν, μετά στον κύριο Τούρμες ή και ανάποδα, όπως θέλει. Αλλά πρέπει να προλάβουμε. Κομισιόν, σας ανακοινώνω ήδη από τώρα ότι υπάρχουν ακόμα ερωτήματα και θα συζητήσουμε και διεξοδικότερα μαζί σας άλλη περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μπορείτε να είστε σύντομοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Στόχος μας είναι το 20%. Αυτός είναι ο στόχος που έχουν υιοθετήσει από το 2007 όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Εκεί λοιπόν στοχεύουμε και διατηρούμε το στόχο αυτό. Εκεί χρειάζεται να φτάσουμε. Συμφωνούμε ότι υπάρχει περιθώριο συζητήσεως των ε, λεπτομεριών για παράδειγμα για το 8 ή για το άρθρο 6 όπως είπε η κυρία Χόλ κλπ. Το να απαντήσω σε όλα τα σχόλια που ακούστηκαν είναι δυνατόν. Θα επιλέξω ένα ή δύο. Απατώντας τον κύριο Βιδάλ Κουάδρας για την συμπαραγωγή, αξίζει το κόπο να τονιστεί ότι αν και είναι διαφορετικές οι ανάγκες, ακόμα και πόλεις όπως η Βαρκελόνη κάνει τώρα μια μεγάλη επέκταση της ε, ε, συμπαραγωγής για τη θέρμανση. Δεν είναι λοιπόν μονάχα θέμα των βόρειων περιοχών και τα σύγχρονα συστήματα συμπαραγωγής με δυνατότητα αποθήκευσης της θερμικής ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν καλούς εταίρους. Δεν θέλουμε λοιπόν να μειωθεί το φιλόδοξο των στόχων προς την κατεύθυνση αυτή. Το ίδιο ο κ. Βιδάλ μίλησε για το άρθρο 6 λέγοντας ότι δεν είναι σωστό οι εναλλακτικέ επιλογές να εξετάζονται πρώτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο λόγος για τον οποίο κάναμε τη σχετική πρόταση είναι διότι για τις υποχρεώσεις ενεργειακής αποδοτικότητας υπάρχουν ξεκάθαρες απαιτήσει και του επίπεδου και της επαλήθευση, και της μη αντιστρεψιμότητας. Εάν υπήρχαν διάφορες επιλογές στο κείμενο δεν θα λέγαμε ότι ε, δεν θα επιμέναμε ότι υπάρχει ανάγκη ε, επαλήθευσης εξάντε. Τέλος υπάρχει ένας αριθμός θεμάτων σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη. Για τους κυρίους Κουάδρας και Κάρινς θα πω ότι οι μελέτες επιπτώσεων μας βασίζονται στην συνέχιση και μάλιστα και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης σε μια περίοδο οικονομικών δυσχεριών είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς άλλο τομέα που να είναι σημαντικότερος από την εξοικονόμηση της ενέργειας και για να αποφευθούν οι σπατάλες αλλά και για να κινητοποιηθεί η ανάπτυξη. Μία από τις ερωτήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι πώς μπορούμε να ζητήσουμε από τις τράπεζες να δανείζουν ξανά. Πώς μπορούν πιο συγκεκριμένα οι τράπεζες να αρχίσουν να δίνουν δάνεια για έργα αύξησης της αποδοτικότητας τη ενέργεια. Υπάρχουν λύσεις βέβαια οι οποίες ε, εντάσσονται στην οικονομική μας ατζέντα. Για την μελέτη επιπτώσεων μιλούμε για ε, μέχρι το 2020 θετική, θετικό αντίκτυπο στο ε, ΑΕΠ της τάξης των 34 δις μέχρι το 2020 όπως είπα και ούτω καθεξής. Η κυρία Καλάσκα Παλίνσκα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές εθνικές συνθήκες και για το πώς θα εξυπηρετήσουμε τους στόχους. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακριβώς ζητούμε από κάθε χώρα μέλος να θέσει δικούς της εθνικούς στόχους. Αυτοί οι στόχοι ε, εμφανίζονται ως απόλυτη κατανάλωση ενέργειας. Όμως στην πρότασή μας κάθε χώρα μέλος έχει τη δυνατότητα να ε, κάνει δικές της προτάσεις και μόνο εάν οι προτάσεις αυτές δεν φτάνουν το 20% μπορούμε να επανέλθουμε με κατάθεση προτάσεως δεσμευτικών στόχων. Η κυρία Τελικαστήγιο, να μια στιγμή να πω ακόμη στην κυρία Παλίνσκα, ότι δεν υπάρχει ανάγκη να εκφράζονται οι, ε, οι στόχοι σε, με όρους έντασης της ενέργειας. Η κυρία Δερκαστήριο είπε να μείνουμε, αν μείνουμε σε αυτή την προσέγγιση χάνουμε τότε τα δεσμευτικά μέτρα. Για την ώρα ωστόσο οι χώρες μέλη στοχεύουν στο 14% και όχι στο 20% της εξοικονόμησης. Αν θέλουμε λοιπόν όμως δεσμευτικούς στόχους τότε χρειαζόμαστε και δεσμευτικά μέτρα. Κάποιο από τα δύο μας χρειάζεται για να επανέλθουμε στην πορεία προς το στόχο του 20%. Θα αρκεστώ σε αυτά για την ώρα και θα περιμένω την συνέχεια της συζητήσεως. Κλοντ Τούρμες. Δεν είμαι σε θέση να περάσω στις λεπτομέρειες σε όλα τα θέματα. Θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε συγκεκριμένα βασικά θέματα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας στη συζήτηση. Αυτά τα οποία είπε η κυρία Δεκαστήγιο δείχνουν το δίλημα στο οποίο βρισκόμαστε. Σε αυτή τη φάση οι κυβερνήσεις αρνούνται δεσμευτικούς στόχους και έτσι μας αναγκάζουν να προτείνουμε νέα μέτρα. Αυτό το οποίο θα κάνω με τρεπολογίες είναι να προτείνω σε ένα πίνακα τους συγκεκριμένους πρωτογενείς ενεργειακούς στόχους που ζήτησε η κυρία Ντελκαστήγιο. Και εδώ έχουμε και εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας, θα δούμε αν οι κυβερνήσεις τελικά τότε ε, ε, θεωρήσουν ότι είναι σοβαροί οι δυνατότητες να θέσουν, να δημιουργήσουν εθνικούς στόχους. Εγώ δεν μπορώ να θέσω συγκεκριμένους στόχους σήμερα, αλλά να πούνε οι κυβερνήσεις ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους επιθυμούν ποσοτικά. Τώρα για τις γενικές ιδέες, για το ποιους δείκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Σαν παράδειγμα, η εντατικότητα της ενέργειας ανά ΑΕΠ. Δεν είναι καλό αυτό. Γιατί στην ουσία διώχνεις από μια οικονομία ας πούμε τρία χαλιβουργία, τα αντικαθιστάς από δύο τράπεζες, Οπότε σε αυτή την περίπτωση αυξάνει το ΑΕΠ σου ή το κρατά το ίδιο και έχει μείωση τη ενέργεια. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό όμω. Οι δείκτε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 368 και οι προβολές, <clears throat> οι χονδρικέ προβολές οι οποίες γίνονται σε σχέση με την αναφορά με τους πρωτογενείς στόχους ενέργειας παρουσιάζει πλέον γιατί μας δίνει κάποιες κατευθύνσεις που βαδίζει μια χώρα και τι πρωτογενή ενέργεια έχει στη διάθεσή της σε επίπεδο υποδομών. Αν δεν έχουμε από την άλλη συγκεκριμένες μετρήσιμες ποσότητες, δεν θα ξέρει κανείς πού, πού θα πρέπει να επενδύσει. Το input και το output, σαν παράδειγμα το ίδιο και στην χαλιβουργία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι θετικό για να θέσει κανείς στόχους, αλλά ο χάλιβας σαν παράδειγμα δεν είναι ένας, υπάρχουν 150 διαφορετικά είδη και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη μία παραγωγή με την άλλη. Λοιπόν, το θέμα της έντασης της ενέργειας, μια ιδέα στην οποία προωθούν πάρα πολλά λόμπι, δεν έχει μέλλον. Δεν έχει μέλλον γιατί δεν θα μας οδηγήσει σε τίποτα το οποίο να μοιάζει με χρήσιμο δίκτυ. Θα πρέπει ίσως να ετοιμάσω ένα σύντομο κείμενο εξηγώντα τι είναι οι στόχοι τους οποίους επιθυμούμε, ποιοι είναι οι δείκτες που θα περιλαμβάνουν και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε. Το θέμα του 3% στην επιφάνεια των κτηρίων τώρα. Το 3% σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν 33 χρόνια για να ανακαινήσουν τα κτίρια τους συνολικά. Από το 2014 και μετά, δηλαδή το 2047 θα πρέπει να έχουν φέρει εις πέρα στις αλλαγές. Τώρα αυτό το θεωρείται υπερφιλόδοξο. Δηλαδή όλα τα κτίρια που ελέγχουν οι τοπικές και οι εθνικές αρχές να ανακαινιστούν μέχρι το 2047 θεωρείται ότι είναι υπερβολικό. Εγώ δεν μπορώ να βρω ένα άλλο μέτρο από την επιφάνεια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο σαν στόχος. Για το άρθρο 6. Χαίρομαι γιατί υπάρχει αρκετή υποστήριξη για το 1,5%. Η παρατήρηση την οποία έκανε ο κύριος Πίπερ για τους βιοτέχνες. Και εγώ είχα αντιπροσωπεία με την Ομοσπονδία, εν περιπτώσει, και είδα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έγιναν κάποιες αξιολογήσεις σε σχέση με τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας από τις μικρές επιχειρήσεις. Και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο θα χτυπήσει ε, τις μικρές εταιρείες. Και νομίζω ότι μικρά καταστήματα και μικρές επιχειρήσεις γενικά και στον τομέα της μόνωσης μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά πράγματα εύκολα. Κοιτάξτε, θα μας εγκαταλείψουν οι διευμηνείς. Δύο λεπτά τελειώνω στην αγγλική, έτσι και αλλιώς οι περισσότεροι από μας. Δύο λεπτά τελειώνω, λέει ο κύριος Τούρμες. Για το άρθρο 10, για την παραγωγή ενέργειας και θέρμανσης μαζί. Είναι μια πρόκληση αυτό που έθεσα. Το θέμα είναι να δούμε ποια είναι τα κριτήρια για τις αναλύσεις κόστους-οφέλους. Κάθε εταιρεία αν είναι ανεξάρτητη να πάρει τα μέτρα δεν θα πάρει κανένα μέτρο. Η κυβέρνηση της Δανίας καθόρισε τα κριτήρια για τον καθορισμό του τι είναι αποτελεσματικό σε επίπεδο κόστους και τι δεν είναι. Αν δεν τα καθορίσεις τότε σε αυτή την περίπτωση ανοίγεις την πόρτα για παρανομίες και εξαιρέσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε μια συζήτηση για τα κριτήρια για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής. Γι' αυτά που είπε ο κύριος Πρόβερα για τα κτίρια ιστορικού χαρακτήρα. Κοιτάξτε, σας προτείνω να καταθέσετε μία τροπολογία για να διευκρινίσετε ακριβώς τι πρέπει να γίνει και σε σχέση με την οδηγία με τα κτίρια. Το 3% δεν αφορά τα ιστορικά κτίρια. Πολλές φορές η νομοθεσία είναι πάρα πολύ περίπλοκη και πρέπει να την απλουστεύσουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να το διευκρινίσετε. Αυτό νομίζω θα είναι καλό για όλους. Και τέλος, Έχετε δίκιο. Το θέμα απαιτεί πολιτιστική αλλαγή, απαιτεί εμπλοκή των πολιτών, απαιτεί την κατάρτιση των βιοτεχνών, απαιτεί την σωστή ενημέρωση των καταναλωτών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα πρόγραμμα εμπλοκής από τα κάτω προς τα άνω όλων των ενδιαφερομένων. Έτσι θα πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει περισσότερα χρήματα. Τότε μόνο οι τοπικές αρχές, ε, ε, η εκπροσώπηση των καταναλωτών θα μπορέσει να συνεργαστούν όλοι αυτοί μαζί μας για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα στην ενέργεια. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στη διάθεσή σας στο Στρασβούργο. Μπορούμε να έχουμε τέτα τέτ συναντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη διερμηνία. Θα δούμε τι θα κάνουμε την άλλη φορά. 7 Νοεμβρίου η κατάθεση προθεσμίας των απολογιών.